Good afternoon. Back to work. are resuming. Καλησπέρα. Συνεχίζουμε τις εργασίες ε, της συνεδρίασης της Επιτροπής Ελευθεριών με το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. Ο κύριος Ρόουντ, συνάδελφος, είναι ο εισηγητής και το ζήτημα εδώ είναι μια πρόταση κανονισμού για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στις 15 Απριλίου ε, προέβησε μια ανταλλαγή απόψεων. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης Πρώτα θα μας μιλήσει ο εισηγητής ο κύριος Ρόουντ και στη συνέχεια θα έχουμε συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το γεγονός ότι αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υφιστάμενης οδηγίας όχι μόνο μέσω επέκτασης του νομικού πλαισίου αλλά και μέσω της εισαγωγής αυξανόμενης ε, ασφάλειας δικαίου. Είναι ένα πολύ απαραίτητο βήμα για μια ε, ομαλώς λειτουργούσα εσωτερική αγορά που θα διευκολύνει τους καταναλωτές και τις εταιρείες ε, να προβαίνουν σε διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές και να έχουν και ταχύτερες συναλλαγές. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω την υποστήριξή μου προς τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξετάσει τις διάφορες πτυχές της, ε, της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω ισχυρότερων μηχανισμών αμοιβέ αναγνώρισης. Ωστόσο, δεν έχουμε εδώ ένα μοντέλο το οποίο εξασφαλίζει επαρκή ασφάλεια με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες. Η κύρια αιστεία του σχέδιου γνωμοδότησής μου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των ε, ηλεκτρονικών συναλλαγών και της ασφάλειας των συναλλαγών και να αντιμετωπίσω τις ασάφειες και τις ε, αδυναμίες του κοινωνισμού στην πράξη. Υπάρχει το σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης η γνωμοδότηση προσπαθεί να μειώσει την περιττή γραφειοκρατία και να ενισχύσει το ρόλο εταιριών και κρατών μελών και να υπάρχει και ένα σαφής συντονιστικός μηχανισμός. Η γνωμοδότηση επίσης ασχολείται με το θέμα της ευθύνης το οποίο νομίζω έχει έναν πολύ ευρύ ορισμό στην πρόταση της Επιτροπής και θα μπορούσε να δημιουργήσει περιτά εμπόδια στην ανάπτυξη του ψηφιακού τομέα όπως σε μια πρόσφατη συνάντηση με τους σκιώδες εισηγητές ε, υπό το φως των πρόσφατων ανταλλαγών απόψεων αποφάσισα να ασχοληθώ και με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, μάλλον να μην μιλήσω για την προστασία των προσωπικών δεδομένων γιατί αυτά θα αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο άλλης, ε, άλλης πρωτοβουλίας. Από ό,τι καταλαβαίνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το, το σύστημα, τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης καλύπτονται ανεπαρκώς και εμέσως μόνο από την υφιστάμενη πρόταση. Ωστόσο, είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλω να συζητήσω και μαζί σας, αλλά παραμένω ανοιχτός στη δυνατότητα να υποβάλουμε μια τροπολογία πριν από την, ε, τις 6 Ιουνίου που είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης. Και να δούμε τώρα εάν θέλουν τα... οι ευρωβουλευτές να λάβουν μέρος στη συζήτηση. Η κυρία Γκυγιώμα, πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματος κυρία Σέτ που είναι σκιώδης ε, για αυτό το ζήτημα. Δεν μπορεί όμως να έρθει σήμερα και επειδή δεν είμαστε πολύ άριθμοι και μου έχει στείλει και τις παρατηρήσεις στα αγγλικά, θα συνεχίσω στα αγγλικά. Καλώς ορίζω την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλό εφαλτήριο και στηρίζουμε τις προσπάθειες για να έχουμε συγκρότηση νομικού πλαισίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση, Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον κανονισμό όμως δεν είναι σαφής κατά τη γνώμη της και δεν εξυπηρετεί τους στόχους ούτε το, επιθυμητό περιεχόμενο. Υποστηρίζει την έκθεση ε, με στόχο να μειωθεί ο αριθμός των κατεξουσιοδότηση υπεράξεων για να έχει μεγαλύτερο περιθώριο λιγμών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη γενικότερη προσέγγιση του εισηγητή επίση, για την προσπάθεια δημιουργία διαλειτουργικότητας, ενώ ταυτόχρονα σεβόμαστε όμω τι εθνικέ προσεγγίσεις. Η τεχνική διαλειτουργικότητα θα έπρεπε στο μέτρο του δυνατού να είναι τεχνολογικά ουδέτερη με τρόπο ώστε οι μεθοδολογίες των κρατών μελών να γίνουν σεβαστές. Χρειαζόμαστε ισορροπία ανάμεσα στο επίπεδο ασφαλείας που χρειαζόμαστε για να υπάρχει αποδοχή από τους πολίτες Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκή Ένωση για να το εξορροπήσουμε με το κόστος και τις υπόλοιπε συνέπειε ε, από την πλευρά των παρόχων. Ε, από αυτή την πλευρά θα πρέπει επίσης ε, να θέσουμε το θέμα της ανάληψης ευθύνης και της απόδοσης ευθύνης όπως βλέπουμε στο σχέδιο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να εξετάσει εντελεχέστερα την πρόταση για να δει αν επιτυγχάνεται αυτή η ισορροπία. Τέλος, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που ε, θα προσφέρονται στα πλαίσια αυτού του κανονισμού θα πρέπει να καλύπτουν και τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Η συμμετοχή τους στην ψηφιακή ενιαία αγορά ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε όλους τους επιμέρους τομείς και θα καταθέσει σχετικές τροπολογίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Λόπε Αγγιλάρη, σας ευχαριστούμε κυρία Γιγιόμ που παρουσιάσατε την άψο της κυρίας σεχέζε με την ιδιότητα της σκιώδους της ηγήτριας, ο κύριος Σεντός Χέντε. Κύριε Σεντών, σας ακούμε. Ως σκιώδης του ΕΛΚ θα ήθελα να κάνω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, θέλουμε να ε, θεσπιστεί κανονισμός και όχι οδηγία. Το σχέδιο του κυρίου Ρόντ προσφέρει το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας ε, που δεν παράσχει, παρέχει συγγνώμη, ο κανονισμός. Σε σχέση με την προστασία των δεδομένων, η οδηγία θα πρέπει να καλύψει και προγράμματα ταυτοποίησης για να καλυφθούν οι ανάγκες των υποπτικών οργάνων. Ε, το άρθρο 11 ως εκ τούτου θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί επακριβέστερα, διότι ε, η επεξεργασία των δεδομένων από τους παρόχους θα πρέπει να υπάρχει στις διατάξεις αυτού του άρθρου. Βάζει το άρθρο 13 τώρα και οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τον στόχο της συλλογή των προσωπικών τους δεδομένων. Συμφωνώ με τον εισηγητή, τον κύριο Ρόντε, δηλαδή θα πρέπει να ορίσουμε επακριβέστερα τα επίπεδα ασφαλείας μέσα στον κανονισμό για να μην υπάρξουν αμφισημίες. Ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο χρήσης ε, πράξεων κατεξουσιοδότησης ε, και, εφαρμοστικών, και το ρόλο των εφαρμοστικών πράξεων σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι του κανονισμού. Ένας ισχυρός μηχανισμός αμοιβαίας αναγνώρισης ανάμεσα στα διάφορα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης ανακράτως μέλος έχει κέρια σημασία αυτό καλύπτει έναν μηχανισμό συντονισμού αλλά και εποπτείας ε, που ε, θα ελαφρύνει το άχθος ε, και των παρόχων αλλά και των επιχειρήσεων. Τέλος, Τονίζω ότι τα επίπεδα ασφάλειας για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις και τις ηλεκτρονικές υπογραφές θα πρέπει να ενισχυθεί για να αναβαθμιστεί και η ασφάλεια δικαίου ε, ε, από πλευράς μου θα καταθέσω τροπολογίες ε, για να ενισχύσω το έργο του κυρίου Ρόντ. Σας ευχαριστώ. Άλμπρεχτ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Ρόντε για τη δουλειά που έχει κάνει. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό σημείο, ιδίως όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Και το πιο σημαντικό είναι η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση όσον αφορά τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης. Έχω ακόμη κάποιες αμφιβολίες για τη διασύνδεση μεταξύ αυτών των τομέων που ρυθμίζουμε εδώ. Καλό θα ήταν λοιπόν στον κανονισμό να το διευκρινίσουμε περισσότερο. Και όσον αφορά την ασφάλεια δικαίου, επίσης θα ήταν χρήσιμο να γίνει αυτή η διευκρίνηση. Όσον αφορά τα θέματα προστασίας δεδομένων, καλό θα ήταν να παραπέμπουμε στο Γενικό Κανονισμό για την προστασία δεδομένων και τους ίδιους κανόνες να εφαρμόσουμε και εδώ. Τους ίδιους κανονισμούς που έχουμε στον Γενικό Κανονισμό. Ευχαριστώ. Κύριε Μπρόνς, δεν σας είχα δει. Ναι, ευχαριστώ. Κάθε προσπάθεια που έχω κάνει να αγοράσω κάτι ψηφιακά ε, απέτυχε και ίσως να είναι κάπως αφελής η παρέμβασή μου. όταν μιλάμε για νομοθεσία, καλό θα ήταν να υιοθετήσουμε μια προσέγγιση ε, εξέτασης της τωρινής κατάστασης, να δούμε τι πήγε στραβά μέχρι τώρα, τι προβλήματα προέκυψαν και απαιτείται αυτή η νομοθεσία. Το πρόβλημα είναι η απάτη, η προσπάθεια απάτης στην προσπάθεια αγοράς ή ε, εμπορευμάτων στο όνομα κάποιου άλλου. Ε, υπήρχαν κάποιες διατάξεις για ρύθμιση, υπάρχει νομοθεσία και τι είδους νομοθεσία. Έχουμε κάποια ε, παραδείγματα παραβίασης της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων. Ευχαριστούμε κύριε Μπρόνς για τα σχόλιά σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Προεδρία του Συμβουλίου, η Επιτροπή καταρχήν. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τα μέλη της Επιτροπής που έλαβαν το λόγο υπέρ των προτάσεων της Επιτροπής και θα ήθελα να υποφεληθώ της ευκαιρίας για να τονίσω ότι όντως και εμείς έχουμε τις ίδιες ανησυχίες όπως αυτές που εκφράστηκαν από τον εισηγητή. Θέλουμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε το επαρκές επίπεδο προστασίας για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και να διασφαλίσουμε ότι η προστασία δεδομένων θα ισχύσει για όλους ε, τους εμπλεκομένους. Και αυτό έχει και σχέση με τη μεταρρύθμιση του τωρινού πλαισίου για την προστασία δεδομένων για τους παρόχους υπηρεσιών ε, θεωρήσαμε ότι είναι σκόπιμο να έχουμε συγκεκριμένες διατάξεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ε, οι φορείς της αγοράς και πώς διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα. Τέλος, ε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η πρόθεσή μας είναι να έχουμε πρότυπα που θα επιτρέπουν τεχνική διαλειτουργικότητα και ουδετερότητα. Και αυτό προσπαθήσαμε να το θέσουμε στον πυρήνα της πρότασης αυτής. Δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να απαντήσω και στην ερώτηση που έγινε για το τι προβλήματα υπήρξαν μέχρι τώρα. Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω ότι η πρόταση αυτή ξεκίνησε από ένα πρώτο πλαίσιο για την ηλεκτρονική υπογραφή και μόνο και όχι για τις υπηρεσίες που τώρα καλύπτει ο κανονισμός. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι δεν υπήρχε, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα διευκολύνει ε, τα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης για τους πολίτες και για τους καταναλωτές, ώστε να βασίζονται σε τέτοια μέσα και να περιορίζουν τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να δίδουν στους παρόχους υπηρεσιών για ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε μια πρόταση όπως αυτή που τώρα υποβάλλεται. Ευχαριστώ πολύ ε, τον κύριο Σαβίδα, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επανέρχομαι στον εισηγητή. Κύριε Ρόντε, έχετε το λόγο για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα απαντήσω προ τον κύριο Μπρόνς. Ε, η απάντησή μου θα είναι ίδια όπω και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ πλήρω με την απάντηση αυτή. Προ την κυρία Χέτ τώρα και τον κύριο Άλμπρεχτ και τον κύριο Σελβιλάμπα. Και ζητώ συγγνώμη αν προφέρω λάθος το όνομά σα. Θεωρώ ότι είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. όπως είχαμε πει και στις 19 Μαΐου στη συνάντηση και μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες ή σχόλια τα οποία θα λάβουμε υπόψη μας. Η τελική ημερομηνία είναι η 6η Ιουνίου. Θα τα λάβουμε υπόψη και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μία συνάντηση να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες και είμαι σίγουρο ότι θα βρούμε μία κοινή γραμμή. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν δυσκολίες. Είμαι ανοιχτό ε, στις προτάσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τα σχόλιά σας και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Ρόντα, ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες. Το είπατε κι εσείς ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 6η Ιουνίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στις 8 ή στις 9 Ιουλίου. Και τώρα Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Μύρια Βασιλιάδου, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίστρια για θέματα εμπορίου ανθρώπων. Τώρα έρχεται στην αίθουσα και την καλωσορίζουμε. We να καλωσορίσουμε την κυρία Μύρια Βασιλιάδου, συντονίστρια στον Ευρωπαϊκό Φορέα Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπινων Όντων, για να μας ενημερώσει για τις δραστηριότητες, τις σχετικές, καθώς και την έκθεση της Eurostat σχετικά με την εμπορία των ανθρωπίνων όντων. Από το το 2013 εκδόθηκαν δύο σημαντικά κείμενα από την Ευρωπαϊκή Έννοια. Η έκθεση της Eurostart τον Απρίλιο, στις 15 Απριλίου, που τόνισε ότι 23.632 άτομα ε, ταυτοποιήθηκαν ως θύματα εμπορίας ε, ανθρώπινων όντων στην περίοδο 2008-2012 με αυξημένους αριθμούς από το 2008 μέχρι το 2010 και παρόλα αυτά οι καταδίκες μειώθηκαν κατά 30% κατά την ίδια χρονική περίοδο. Δεύτερον, υπάρχει ένας οδηγός για τα ευρωπαϊκά δικαιώματα των θυμάτων της εμπορίας ανθρωπίνων όντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να απαλείψει ε, μεταξύ του 2012 και 2016 την εμπορία ανθρωπίνων όντων. Έχουμε την τιμή να καλωσορίσουμε την κυρία Βασιλιάδου, συντονίστρια, η οποία θα μας πει κάποια παραπάνω για την έκθεση αυτή και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση. Κυρία Βασιλιάδου, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και για το έντονο ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα της εμπορίας των ανθρωπίνων όντων. Νομίζω ότι η απλή αριθμή και μόνο των ε, ερωτήσεων στο Κοινοβούλιο λέει πολλά από μόνος του και δείχνει την υποστήριξη και το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Και για τον λόγο αυτό εξακολουθούμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας απαντούμε επαρκώς και έγκαιρα. Ε, πώς έχει η κατάσταση σήμερα. Ε, είναι η δουλεία της εποχής μας. Είναι κατάφορος, κατάφορη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, απαγορεύεται ρητός από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι μια σοβαρή μορφή εγκλήματος, συχνά οργανωμένου εγκλήματος. Είναι ένα ε, φαινόμενο που αφορά συγκεκριμένο φύλλο και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζετε. Όλες οι πληροφορίες που θα σας δώσω σήμερα βασίζονται πάνω σε αυτά που προανέφερα. Τρία σημεία. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος επειδή υπάρχει πολιτική βούληση ε, και Υπάρχει, έχει αυξηθεί και το σχετικό ενδιαφέρον. Θα μιλήσω καταρχήν για την νομοθεσία, στη συνέχεια για την πολιτική και στη συνέχεια για τη χρηματοδότηση. Όσο αφορά την νομοθεσία, έχουμε την οδηγία του 2011 για την εμπορία των ανθρώπινων όντων. Επρόκειτο να μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο μέχρι τις 6 Απριλίου 2013. Αυτή ήταν η καταληκτική ημερομηνία. Έχουμε αρχίσει ήδη να εξετάσουμε τα μέτρα μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών. Έχουμε διευκολύνει μια άτυπη ομάδα στην οποία συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη και όπου μπορούν να συζητήσουν τη δική τους ερμηνεία των διαφόρων άρθρων της οδηγίας. Κατά αποτέλεσμα, σήμερα εννέα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει πλήρως την οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο. Τέσσερα κράτη-μέλη μας έχουν ενημερώσει για μερική μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο και θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα, όλα τα κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν την οδηγία στο εσωτερικό τους δίκαιο και βασιζόμαστε πάνω στις υπηρεσίες της Επιτροπής να μας βοηθήσουν. Τώρα, χάραξη πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απάλληψη της εμπορίας ανθρωπίνων όντων του 2012 μέχρι το 2016. Υπάρχουν 40 πάρα πολύ φιλόδοξε δράσεις, δεν θα τις παρουσιάσω σήμερα, αλλά θα σας υπενθυμίσω ότι εάν και υπήρξε έντονη υποστήριξη, κυρίως από τον τομέα της κοινωνίας των πολιτών, η Επιτροπή Περιφερειών, η Κοινωνική και Οικονομική Πολιτική και πολλοί άλλοι έχουν δηλώσει την έντονη στήριξή τους για τη δουλειά που κάνουμε. Θα επικεντρωθώ τώρα στην έκθεση της Eurostat, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Ελπίζω να, υπάρχει, να υπάρχουν αντίγραφα, αλλά όχι, όχι, διορθώνει η ομιλήτρια τον εαυτό της. Η έκθεση αυτή έχει ήδη ξεπουληθεί. Έχει εξαντληθεί. Δεν υπάρχουν άλλα αντίγραφα και βρισκόμαστε στη διαδικασία της επανατύπωσης της έκθεσης. Φυσικά μπορείτε να την διαβάσετε ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Σε αυτή την έκθεση της Eurostat για πρώτη φορά έγινε η προσπάθεια να έχουμε στατιστικά στοιχεία για την εμπορία ανθρωπίνων όντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται τα έτη 2008, 2009 και 10. Έχουμε πληροφορίες από τα 27 κράτη-μέλη και από την Κροατία, καθώς και τις χώρες ΣΕΖΕΣ, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Σερβία, Ισλανδία κτλ. Έχουμε επίσης στατιστικά για το συνολικό αριθμό θυμάτων κατά φύλλο, ηλικία και μορφή κακοποίησης, ε, ηθαγένεια, μέτρα προστασίας κτλ. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία ε, περιέχουν πληροφορίες που έχουν δώσει ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ε, υπάρχουν στοιχεία από τις διαδικασίες καταχώρησης στα διάφορα κράτη-μέλη και υπάρχουν και μεταβάσεις δεδομένων. Έχουμε περίπου 23.600 ανθρώπους που έχουν ταυτοποιηθεί ως υποτιθέμενα θύματα για την περίοδο 2008 με 2010. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε όμως είναι ότι αυτή είναι μόνο η κορφή του παγόβουνου φυσικά. Να σας θυμίσω ότι το Διεθνής Οργάνωση Εργασίας για την ίδια περίοδο εκτιμά περίπου 880.000 τα άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που υπήρξαν θύματα καταναγκαστικής εργασίας. Νομίζω πάντα πρέπει να θυμόμαστε καθώς μιλούμε ότι υπάρχουν άντρες, γυναίκες, παιδιά που πολλούνται για σεξ και αναγκαστική εργασία ε, σε, εξαναγκάζονται σε γάμο, ε, χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες ε, κατοίκων ή τα όργανα τους πολλούνται για μεταμοσχεύσεις. Όταν μιλούμε για εμπορία ανθρωπίνων όντων, μιλούμε για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, για κοινωνικό διαρκώς αποκλεισθέντες ανθρώπους, κοινωνικά ευάλωτους και φαίνεται ότι η οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Και γι' αυτό πρέπει να οξύνουμε την προσοχή μας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο αριθμός των θυμάτων εξακριβωμένος ή ανεπιβεβαίωτος έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Αλλά όλο και λιγότεροι έμποροι ανθρωπίνων όντων καταδικάζονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα. Η μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες και νεαρές κοπέλες και το 20% άρενες, 15% επί του συνολικού αριθμού παιδιά. Είναι ένα φαινόμενο που σχετίζεται έντονα με το φύλλο. Ε, σεξουαλική εκμετάλλευση 62%. Οι γυναίκες και οι κοπέλες φυσικά είναι η μεγάλη πλειοψηφία αυτού του ποσοστού και ο αριθμός αυξάνεται. Υπάρχει μια σταθερή άνοδος του ποσοστού σεξουαλικής κακοποίησης. Η εκμετάλλευση για καταναγκαστική εργασία 25% μοιάζει να μειώνεται ο αριθμός όσο αφορά τα επιβεβαιωμένα περιστατικά. Χαίρομαι για αυτή τη μείωση βέβαια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταγράφουμε όσους άρενες απαιτείται στον τομέα της καταναγκαστικής εργασίας, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε την έμφασή μας στη σεξουαλική εκμετάλλευση, νομίζω. Θα, θα σας αποστείλουμε, θα αποστείλουμε και ένα ερωτηματολόγιο. Την επόμενη τριετία θα συνεχίσουμε να συλλέγουμε στοιχεία. Ε, η πρωτοβουλία αυτή έχει τύχη ευνοϊκής ε, υποδοχής. Υπάρχει ένα άλλο παραδοτέο που ελπίζω να έχετε μπροστά σας ή που θα το έχετε μπροστά σας σύντομα. Έχουμε μια δημοσίευση που αφορά τα δικαιώματα των θυμάτων σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο. Όπως είπα και νωρίτερα, η όλη στρατηγική ε, εστιάζεται στα βήματα. Ό,τι κάνουμε εστιάζεται στα θύματα υπάρχει αυτή η δέσμευση. Είμαι περήφανη για αυτή τη δέσμευση και είμαι περήφανη και για αυτή την επισκόπηση αυτής της νομοθεσίας, η οποία παρουσιάζεται με φιλικό προς τον αναγνώστη τρόπο, όλα τα δικαιώματα, πρόσφο, πρόσβαση σε δικαστήρες, σε δικαιοσύνη, σε κοινωνικές υπηρεσίες, σε υπηρεσίες υγείας κτλ. Όλα αυτά τα δίνουμε σε προσβάσιμη γλώσσα το δεύτερο τμήμα του εγγράφου αναφέρει και συγκεκριμένα άρθρα οδηγιών. Αυτό θα υπάρχει σε 23 γλώσσες, θα είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά για να διευκολύνουμε το, τη δουλειά των υπαλλήλων αλλά κυρίως των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για τα θύματα. Η Ιρλανδική Προεδρία θα προάγει τη διάδοση αυτής της δημοσίευσης ε, που θεωρούμε ότι και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όσο αφορά τους συνεργάτες μας, τους πρωταγωνιστές, ε, μερικοί είναι λιγότερο προφανείς φυσικά με την ε, Europol, με την Eurojust, με την Eurofrontex, αλλά και με άλλους φορείς. Και όπως οι επιθεωρητές εργασίας. Πριν από τρεις μέρες είχαμε λάβει μέρος σε μία άτυπη συνάντηση επιθεωρητών εργασίας στο Δουβλίνο και για πρώτη φορά η εμπορία των ανθρωπίνων όντων ήταν μέρος της ημερήσιας διάταξης. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι εργάζονται στον τομέα της απασχόλησης, του δικαίου της απασχόλησης, ε, θα ευαισθητοποιηθούν στο θέμα αυτό. Ένας άλλος ε, συνεργάτης είναι η κοινωνία των πολιτών. Ε, η ιδέα προήλθε από εσάς, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί κάποιοι ευρωβουλευτές αναρωτήθηκαν αν έχουμε κάποιο δίκτυο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των θυμάτων των... της εμπορίας ε, ανθρωπίνων όντων. Υπήρξε πολύ έντονο ενδιαφέρον από τις οργανώσεις ανά την Ευρώπη και ε, είχαμε εκπροσώπους όπως είπα από τα 27 κράτη-μέλη και από την Κροατία και από άλλους. Είναι, ήταν η πρώτη συνάντηση του είδους, στο πλαίσιο της οποίας ε, πολλές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τα θύματα της εμπορίας ανθρωπίων όντων, συγκεντρώθηκαν μαζί, αντάλλαξαν πληροφορίες, ενημερώθηκαν καλύτερα και έτσι μπορούν να συνεισφέρουν καλύτερα στην υλοποίηση της στρατηγικής και της οδηγίας. Είχαμε υφιστάμενα δίκτυα, αλλά ήταν πολύ συγκεκριμένα δίκτυα, περιορισμένα. Θελήσαμε να επεκτείνουμε την εμβέλεια ε, του διαβήματος αυτού για να έχουμε και καλύτερα εργαλεία αντιμετώπισης της κατάστασης. Ε, περισσότερο έχουν συμμετέχει οργανώσεις γυναικών και παιδιών. Θέλω να μιλήσω τώρα για τη διάσταση του φύλου. Εξήγησα ότι το 96% όλων των θυμάτων, ιδίως ε, για τη σεξουαλική κακοποίηση, είναι γυναίκες και νεαρές κοπέλες. Ε, συμπεριλαμβάνεται η εκμετάλλευση της πορνείας στο δρόμο, στις βιτρίνες καταστημάτων, στην πορνογραφία κτλ. Τα στοιχεία τονίζουν τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της βιομηχανίας του σεξ και των δικτύων εμπορίας ανθρωπίνων όντων ή μεταξύ των δικτύων πορνείας και των δικτύων εμπορίας. Θέλουμε να εντείνουμε τη δουλειά μας για την σεξουαλική κακοποίηση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε μόνο σε μία μορφή, στην καταναγκαστική εργασία, για παράδειγμα γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουμε καθόλου περιορίσει τη σεξουαλική κακοποίηση. Τα κράτη-μέλη ε, καλούνται να λάβουν πρακτικά μέτρα για να μειώσουν τη ζήτηση, ρητά ζητείται αυτό από τα κράτη-μέλη, και να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη. Επίσης, να υπάρξουν μέτρα να ενταθεί η ποινική ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων καθώς και η και των χρηστών όταν υπάρχει γνώση ότι το άτομο είναι θύμα εμπορίας ανθρώπινων όντων. Υπάρχει βέβαια η βία κατά των γυναικών, το θέμα αυτό. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέδεσε τα δύο αυτά θέματα και χαίρομαι που τώρα πια θα υπάρχει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτό το είδος της βίας κατά των γυναικών. Μίλησε για τους επιθεωρητές εργασίας ε, και για την κοινωνία των πολιτών. Η άλλη ενδιαφερόμενη πλευρά είναι ο ιδιωτικός τομέας, ο επιχειρηματικός τομέας. Ε, προσπαθούμε σκληρά να υπάρξει μία ένας συνασπισμός επιχειρήσεων μέχρι το 2014 για να δούμε πώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και εταιρείες μπορούν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη επίγνωση, καλύτερο έλεγχο αυτών των πραγμάτων και στις εφοδιαστικές τους αλυσίδες. Μέχρι τις 6 Απριλίου θα πρέπει να θεσπιστούν τα, οι ή τα άτομα που θα αναλάβουν το συντονιστικό ρόλο ε, όλων αυτών των δράσεων και θα υποβάλουν εκθέσεις οι οποίες θα πρέπει να φτάνουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεργαζόμαστε επίσης με υπηρεσίες δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Πριν από δύο χρόνια υπογράφτηκε μια δήλωση ε, από τον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων για συνεργασία με σκοπό την μείωση της εμπορίας ανθρωπινών όντων. Ε, Υπογράφηκε η διακήρυξη αυτή από όλους τους αρμοδίους, ε, τους επιτρόπους και τα λοιπά. Συνεργαζόμαστε μαζί τους, έχουμε τακτικά συναντήσεις για να συντονίσουμε καλύτερα τις εργασίες μας. Συνεργαζόμαστε επίσης με, την, ε, με τον Οργανισμό Θεμελιδιών Δικαιωμάτων, ιδίως για τα παιδιά που είναι θύματα και για να προετοιμάσουμε και ένα εργαλείο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης μέχρι το 2014 στα θέματα εμπορίας ανθρωπίνων όντων. Υπάρχει φυσικά και οι διεθνείς συμβάσεις για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ένα από τα πιο επιτυχημένα εργαλεία του επιχειρησιακού πλάνου που υιοθέτησαν τα κράτη-μέλη. Ε, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη προσήλωση και δέσμευση οι νέοι στρατηγικοί στόχοι θα συζητηθούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους και φυσικά η εμπορία ανθρωπίνων όντων θα αποτελέσει μέρος της ατζέντα. Εσωτερικά συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις δράσεις, συντονίζουμε 17 υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι γενικές διευθύνσεις, οι οποίες συμμετέχουν όλο και περισσότερο, απασχόληση, μετανάστευση, ανάπτυξη, εμπόριο, επιχειρήσεις, ε, δικαιοσύνη, κατάρτιση και φυσικά και η ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Συνεργαζόμαστε με όλους αυτούς πολύ συστηματικά. Συμμετείχαμε επίσης σε ενδοϊπηρεσιακές ε, διαδικασίες διαβούλευσης ε, καθώς και ενημέρωσης για τα προγράμματα χρηματοδότησης. Και θα κλείσω με τη χρηματοδότηση. Φυσικά είναι θεμελιώδης προϋπόθεση. Είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διευκολύνει το έργο που κάνουμε. Έχουμε προσπαθήσει πρώτον να εξασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση αντιστοιχεί καλύτερα στην πολιτική. Να μην δηλαδή χρηματοδοτούνται έτσι αυθαίρετα προγράμματα τα οποία δεν ευθυγραμμίζονται με τον στόχο μας. Από την άλλη πλευρά προσπαθήσαμε να διαφοροποιήσουμε και όλες τις πηγές χρηματοδότησης. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε τετραπλάσιες αιτήσει, από 20, από 20 περάσαμε σε 60 αιτήσει και έχουμε τετραπλάσιο αριθμό ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων και διαφορετικών κατηγοριών μη κυβερνητικών οργανώσεων που υποβάλλουν αιτήσει. Θέλουμε λοιπόν, όπω είπα, να εξασφαλίσουμε ότι η χρηματοδότηση ταιριάζει, ευθυγραμμίζεται με την ε, υλοποίηση της νομοθεσία. Όλα αυτά υπάρχουν σε ειδικό ιστότοπο. Είναι κάτι μοναδικό που καταφέραμε να κάνουμε. Έχουμε φέρει μαζί όλα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την εμπορία ανθρωπίνων όταν από το 2003 μέχρι σήμερα σε ένα συγκεκριμένο ειδικό ιστότοπο, 11 διαφορετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε όλες. Θέλουμε να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία στην ιστοσελίδα μας, τις πηγές χρηματοδότησης, ε, τι ε, δράσεις χρηματοδοτούνται, σε ποια κράτη-μέλη. Για την εξωτερική διάσταση δεν θα επιμείνω σε αυτό, αλλά έχουμε δύο μεγάλα εργαλεία, την σφαιρική προσέγγιση στη μετανάστευση και την κινητικότητα, καθώς και τη δράση κατά της εμπορίας, έναν από τους πυλώνες ε, της ΚΑΜ. Και Επίσης υπάρχει ένα έγγραφο για την εξωτερική δράση της Ένωσης κατά της εμπορίας των ανθρωπίνων όντων. Συγκεκριμένα τώρα τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει για κάποιες χώρες και περιοχές προτεραιότητες πάνω στις οποίες πρέπει να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει την εμπορία. Έχουμε τέσσερις χώρες προτεραιότητες, οι οποίες επιλέγησαν με μεγάλη προσοχή και έγιναν και πολλές συζητήσεις μέχρι να επιλεχθούν οι συγκεκριμένες χώρες, η Αλβανία, η Βραζιλία, η Κίνα, η Δομινικανή ε, Δημοκρατία, το Μαρόκο, η Νιγηρία, η Ρωσία, το Βιετνάμ, η Τουρκία και η Μαλαισία. Ε, συνεργαζόμαστε λοιπόν με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, και με τις αντιπροσωπείες για να δούμε πώς συγκεκριμένα θα δράσουμε και να πώς θα βρούμε και δωρητές, χρηματοδότε. Έχω και πολλά να σας πω ακόμη, αλλά πρέπει να σταματήσω, να σας πω απλώς ότι η ιστοσελίδα μας πριν από τρεις εβδομάδες, ε, μάλλον τον Μάρτιο, είχε 2.000 κλικ ε, μόνο στην πλατφόρμα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Όλα αυτά κατέστησαν δυνατά επειδή υπήρχε και η έντονη στήριξη αυτού του κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ήσασταν ενθουσιώδης και επίσης διεξοδικότατη κατά την παρουσίαση των επιτευγμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Ας αρχίσουμε την συζήτηση. Ε, ο εκπρόσωπος ή η εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Σακυλιάδου, εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το ζήτημα, όχι, όχι. Λοιπόν, ας αρχίσει η συζήτηση τότε. Κυρία Μπάουερ, ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Βασιλιάδου, πολύ καλά τα νέα σας. Ε, όμως μας απογοήτευσαν λίγο τα κακά σας νέα. Και θα αρχίσω με μια σχετική ερώτηση. Πώς εξηγείτε εσείς το εξαιρετικά απογοητευτικό ε, δεδομένο της ε, ελλειπούς μεταφοράς στην ε, οικία νομοθεσία. φαινόταν ότι όλοι είχαν λάβει σοβαρή δέσμευση. Βλέποντας λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα, ε, αποκαρδιωνόμαστε και ακριβώς τι προτίθεστε να κάνετε για αυτό το ζήτημα και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Έπρεπε όντω να ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσεις των κρατών μας ε, γιατί πρόκειται για ένα πραγματικό πρόβλημα. Πέραν αυτού, ποια άλλη λύση υπάρχει τώρα. Ένα επίσης εξίσου ε, απογοητευτικό αριθμητικό στοιχείο που μου δώσατε είναι η αύξηση του αριθμού των παιδιών ε, στο συνολικό αριθμό των θυμάτων. Θα μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο περισσότερο. Κάτι που με δυσαρεστεί ιδιαίτερως είναι ότι στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ευζήν των παιδιών δεν γίνεται καν μία σε αυτό. Έχοντας υπόψη αυτά που μας είπατε για τα δικαιώματα των θυμάτων και τα όσα έχετε δημοσιεύσει σχετικά, ε, νομίζω δεν είναι καινούριο το ζήτημα για τις ε, προσωρινές ε, άδειες ε, διαμονής και η αντίθεση που υπάρχει με την κείμενη νομοθεσία της Ένωσης και ρωτώ τι σκοπεύετε να κάνετε. Γιατί δεν μπορούμε να το δεχτούμε. οι επιθεωρητές εργασίας και ο ρόλος τους είναι πραγματικά μια πολύ καλή ιδέα από πλευρά σας. κυρίως δεδομένης της επιτυχίας που σημειώσατε, δημιουργήσατε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συνεργασία των αρμοδίων εθνικών οργανισμών και σε αυτά τα πλαίσια είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος των επιθεωρήτων εργασίας για τα ζήτημα της καταναγκαστικής εργασίας και της εμπορίας ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα και όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολο είναι να εντοπιστούν ε, τα θύματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Τελευταία παρατήρηση. Σας συγχαίρω που ε, εισαγαγείται αυτό το ζήτημα στη, στα πλαίσια της αναπτυξιακής πολιτικής, γιατί έτσι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, ούτω ώστε να είναι πιο συνεκτική η πολιτική της Ένωσης. Ε, σας ευχαριστούμε. Ε, Head, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Μπάουερ η κυρία Μπάουερ είπε πολλά από αυτά που είχα και εγώ στο μυαλό μου. Είναι ε, λυπηρά τα ε, στατιστικά δεδομένα που μας δώσατε και κυρίως μας λείπει το, το ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν μεταφέρει στην ε, νομοθεσία τους της Διατάξης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα μπορούσε να στείλει μια σχετική επιστολή στο Συμβούλιο ή να εξετάσουμε κάποια κάποιον άλλο τρόπο για να δείξουμε ότι από ε, πλευράς μας θα πρέπει, θεωρούμε ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση για την εφαρμογή αυτής της τόσο σημαντικής ε, νομοθεσίας. Ε, είναι αυξανόμενα τα νούμερα στην διασυνοριακή εγκληματικότητα και στην Επιτροπή ΚΡΙΜ ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, πώς ακριβώς να αντιμετωπιστεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε αυτό της εμπορίας ανθρώπων. Ε, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και κυρίως να αναλάβουμε περαιτέρω δράση. Είναι εξαιρετική, εξαιρετική η δουλειά που κάνετε και σας συγχαίρουμε. Είναι πάρα πολύ καλό που έχετε ε, πλέον αυτή την πλατφόρμα ε, και παρόλα αυτά τα αρνητικά στατιστικά στοιχεία, η γενικότερη εντύπωση που μας μεταδώσατε είναι θετική και χαίρομαι πάρα πολύ που ε, ασχολείται πισταμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό το ζήτημα. Καλή τύχη σας ευχόμαστε για τη μελλοντική δουλειά σας. Είμαστε πίσω, θα σας υποστηρίξουμε ε, για αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστούμε κυρία Τσέροκά. Κυρία Γιάροκά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και ε, για τις πλέον πρόσφατες ειδήσει που μας κοινοποίησατε. Ε, χαίρομαι για την εμπειρία που έχετε στον τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων και πιστεύω ότι είναι σημαντικό ε, να έχουμε ε, συνεισφορές και από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και από τις τελευταίες επιστημονικές γνώσεις κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας. Και εγώ ίδια είμαι ανθρωπολόγος και όταν ετοιμάζαμε ένα φάκελο για την Βελγική Βουλή, για την επαιτία και το, την εξαναγκασμένη επαιτία και το εμπόριο ανθρώπων, χρησιμοποίησαμε επιστημονική έρευνα ψυχολόγων ε, και αντίστοιχα επιχειρήματα για να βασίσουμε την έκθεσή μας σε σχέση με τη θυματοποίηση των επετών. Πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει αλληλοϊποστήριξη γιατί χωρίς τη δική σας συμμετοχή δεν ακούγονται οι φωνές αυτών που πρέπει να ακουστούν. Και η ανθρωπολογική έρευνα ξέρω ότι δεν χρησιμοποιείται στο βαθμό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει εξαιρετικό υλικό. Και για τα δικαιώματα των παιδιών υπάρχουν ε, στοιχεία και είναι πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης, Χαίρομαι γιατί μιλήσατε για τις εξωτερικές δράσεις που αναλαμβάνετε και για όλες τις ανταλλαγές ε, που γίνονται στο πλαίσιο της Επιτροπής. Ήμουν εισηγήτρια για ένα θέμα που είχε άμεσα σχέση με το εμπόριο ανθρώπων από πολύ απομακρυσμένες περιοχές που πλήττονται από την φτώχεια, ιδίως λόγω της κρίσης σήμερα. Τα θύματα λοιπόν της εμπορίας προέρχονται πολύ συχνά από τέτοιες περιοχές, από μακρισμένες φτωχές περιοχές. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκείται κριτική για το γενικό πλαίσιο και συντάσσονται συστάσεις από την Επιτροπή για την αναθεώρηση του πλαισίου και η δική σας συνεισφορά θα είναι πολύ χρήσιμη. Θέλουμε λοιπόν να έρχεστε στο Κοινοβούλιο και να ενημερώνετε και για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να σας ζητήσω τη γνώμη σας και για το εξής. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έρχομαι από την Ουγγαρία και η μεταφορά σε εθνικό δίκαιο στην Ουγγαρία έχει γίνει πολύ καλά. Αλλά ε, προσπάθησα στην Βελγική ε, Βουλή να ακούσω τι γίνεται για το θέμα αυτό της επαιτίας συγκεκριμένα και των παιδιών επαιτών περισσότερο. Η θέση μου είναι ότι θα πρέπει να απαγορεύεται η επαιτία γιατί αυτό παραβιάζει τα δικαιώματα των παιδιών. Από την άλλη πλευρά, ως ε, ανθρωπολόγος ε, και από την οπτική γωνία των Ρωμά, είναι πολύ χρήσιμο να ακούσουμε τις απόψεις ε, αυτών που δουλεύουν και με τους Ρωμά και μεγαλύτερων μη κυβερνητικών οργανώσεων που ισχυρίζονται ότι είναι δικαίωμα των γονέων και είναι και ένα είδος πολιτιστικής κληρονομιάς. Τέτοιου είδους επιχειρήματα είναι παραπλανητικά πιστεύω. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω τη δική σας γνώμη από αυτού για τα θέματα των Ρωμά. Γιατί ήδη στην Επιτροπή βοηθούν ε, μια ομάδα 120 ε, ακαδημαϊκών για την ε, αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων και για τη χάραξη πολιτικής για αυτό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν και τη δική σας γνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Ρομπέρτα Λόπες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κυρία Βασιλιάδου, για την έκθεσή σας. Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα συνεχίσουμε να επιτυχάνουμε πρόοδους για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω κάποιες διευκρινήσεις. Υπάρχει νομίζω μία σύγχυση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εκμετάλλευσης ε, για εργασία. Η σεξουαλική εκμετάλλευση δεν είναι το ίδιο όπως ε, η εκμετάλλευση για σκοπούς εργασίας. Και αν ε, αναμειγνύουμε τα δύο αυτά θέματα, μπορεί να αποδίδουμε ίδια σημασία και στα δύο. Έχουν μεν σχέση, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η εκμετάλλευση για την εργασία θα μπορούσε να ισχύσει σε οποιονδήποτε έρχεται παράνομα στην αγορά εργασίας μέσω δικτύων εμπορίας, αλλά δεν είναι ίδια τα στοιχεία με αυτά τα οποία βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε πολύ υψηλότερα στοιχεία από τα στοιχεία της έκθεσης. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι πολύ ακριβές αυτό το οποίο συζητάμε στην ε, εκμετάλλευση για σκοπούς εργασίας ε, και ε, εκμετάλλευση και σεξουαλική εκμετάλλευση. Αν επεκτείνουμε αυτό το φαινόμενο ώστε να συμπεριλαμβάνεται και η εκμετάλλευση για εργασία και η σεξουαλική εκμετάλλευση στη σεξουαλική εκμετάλλευση μιλάμε κυρίως για γυναίκες αλλά και για άνδρες και για παιδιά. Πάντως μιλάμε για ομάδες που είναι ευάλωτες και που εξαρτώνται από τα δίκτυα εμπορίας και υπόκειται σε μεγαλύτερους κινδύνους. Γι' αυτό θα πρέπει να καταγγέλλονται ε, τα δίκτυα, αλλά για τα άτομα αυτά είναι δύσκολο να φεύγουν, να βγαίνουν από τα δίκτυα, γιατί είναι εξαρτημένα και ε, ε, είναι πολύ δύσκολο να βγουν από αυτά τα δίκτυα καταγγέλλοντά τα. Πρέπει λοιπόν στην έκθεσή μας να, καταγγέλουμε, να ε, κάνουμε σαφή τη διαφορά μεταξύ εκμετάλλευσης για εργασία και σεξουαλική εκμετάλλευσης, προσδιορίζοντα τι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο. Και έχω και μία ερώτηση. Στην Ισπανία έχει μεταφερθεί σε εθνικό δίκαιο η οδηγία και έχω μάλιστα και τη σχετική έκθεση και βλέπω τα αριθμητικά στοιχεία για την Ισπανία που μου κάνουν εντύπωση. Φαίνεται μια μεγάλη αύξηση από το 2009-2010, αύξηση του αριθμού των θυμάτων. Τετραπλασιάζεται ο αριθμός, πράγμα το οποίο δεν παρατηρείται σε καμία άλλη χώρα. Μια πολύ έντονη αύξηση στα θύματα εμπορίας. Βλέποντας τα δίκτυα εμπορίας από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ε, τους διακινητές που είναι αντικείμενο δίωξης στην Ισπανία, περίπου 300 ε, βλέπω. 300 δίκτυα, 300 διακινητές, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για καταδίκη αυτών. Ίσως η Ισπανία να μην έδωσε καν στοιχεία ως απάντηση. Φαντάζομαι λοιπόν ότι κάποιες χώρες δεν θα έδωσαν στατιστικά στοιχεία. Αλλά από τα μέσα ενημέρωση στην Ισπανία έχουμε πληροφορηθεί πρόσφατα ότι καταδικάστηκαν εννέα άτομα ακριβώς για αυτό το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων. Ίσως ε, οι γυναίκες που είναι αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης στα δίκτυα πορνείας να μην καταγγέλουν τους διακινητές. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε σχετικά στοιχεία, αν έχετε κάποιες πληροφορίες για το αν κάποιες χώρες έχουν δώσει στοιχεία και άλλες χώρες δεν έχουν δώσει στοιχεία για τις καταδίκες. Όσον αφορά τη στρατηγική της Επιτροπής, Δεν υπάρχουν στοιχεία σε όλες τις εκθέσεις. Ε, καλό θα ήταν να δίδεται κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς στα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, να έχουν ένα προστατευόμενο καθεστώς. Οπότε αν αισθάνονται ότι προστατεύονται, θα μπορούν πιο εύκολα να καταγγέλουν τους διακινητές. Είναι μια μορφή υποστήριξης που πρέπει να δώσουμε για να μην διαιωνίζεται αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόνς. Η λέξη εμπορία ετοιμολογικά συνδέεται με την μεταφορά ανθρώπων, κυρίως διαμεθοριακά. Αν δείτε τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών που βλέπω σε αυτό το ενημερωτικό σημείο με τις 15 Απριλίου της Επιτροπής Σημείωμα αναφέρεται σε ανθρώπους που ε, είτε συλλέγονται, είτε μεταφέρονται, είτε διακινούνται μέσω δικτύων με σκοπό την πορνεία. Επειδή ε, χρησιμοποιείται το διαζευτικό «ή», ε, είναι σαν να μπαίνουν σε αυτόν τον ορισμό ε, τα, οι κοπέλες που είναι αντικείμενο πορνείας ακόμη και αν δεν υπάρχει μετακίνηση μέσα στον ορισμό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει τέτοιου είδους διακίνηση μέσα σε τέτοιες ομάδες ε, πληθυσμού από τη μία πόλη στην άλλη. Ε, και τα θύματα και οι θύτες προέρχονται από διαφορετικές ομάδες πληθυσμού. Η πολιτική και η αστυνομία επί χρόνια αρνούνται την ύπαρξη του προβλήματος και μάλιστα απειλούν πολλές φορές αυτούς που λένε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τους απειλούν ότι θα τους διώξουν ποινικά. Ακόμη και ένας πρώην συνάδελφος στο Κοινοβούλιο διώχθηκε ανεπιτυχώς διότι επέστησε την προσοχή του κοινού σε αυτά τα θέματα. πολλά θύματα και πολλά ανήλικα θύματα ακόμη και 13 ετών μένουν έρμεα της τύχης τους λόγω ακριβώς αυτής της πολιτικής. Και ο τρέχον βουλευτής Κίθλι και Γιόρξερ είναι ένα από τα λαμπρά παραδείγματα που το 2006 αρνήθηκε ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ε, τώρα ε, εκμεταλλεύεται αυτό το θέμα ε, υποκρινόμενος ότι ανησυχεί. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα λοιπόν ε, της, ε, ε, της εμπορίας κοριτσιών και αγοριών διεθνώς, αλλά μην ξεχνάμε και άλλες μορφές του ιδίου εγκλήματος. Ευχαριστώ. Κυρία Γκυγιόμ. Ε, ναι, πολλές, πολλές ερωτήσεις ακούσαμε ήδη και θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπε και ο κύριος Δεμένο Λόπες ε, για τη σχέση ανάμεσα ε, στα θύματα, θύματα που ταυτοποιούνται βάσει των στοιχείων που μας κοινοποιήσατε. Μας μιλήσατε για αύξηση 18% σε τρία χρόνια και ταυτόχρονα μας, είπε ότι, μας είπατε ότι έχει μειωθεί ο αριθμός ε, των ε, καταδικών. Ε, χωρίς να μπείτε σε πολλές λεπτομέρειες θα μπορούσατε να επανέλθετε στο, στις καταδίκες και γιατί έχουν μειωθεί ενώ αυξάνεται το αριθμό των θυμάτων. Ε, Ω προ τα στατιστικά στοιχεία, συγγνώμη που επανέρχομαι, αλλά νομίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον. Έχετε μήπω συμπληρωματικά στοιχεία για τις ε, πολιτικές που ακολουθούνται, ε, για την αποκατάσταση των ε, θυμάτων, για το πώς μπορούν στη συνέχεια να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Αν έχετε επιπρόσθετες πληροφορίες, αυτό θα θέλαμε να μάθουμε. Ο κύριος Τρενταφυλλίδης, παρακαλώ. Ε, πολύ σύντομη θα είναι η παρέμβασή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Βασιλιάδου. Ήταν ε, πολύ καλή η παρουσίαση που μας έκανε και να την ευχαριστήσω επίσης και για όλες τις προσπάθειες που καταβάλει. Ήθελα να τη συγχαρώ για τις προσπάθειες αυτές, διότι αποπειράται να αντιμετωπίσει αυτό το φρικιαστικό πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε. Κυρία Βασιλιάδου, Αναφερθήκατε σε διάφορες μορφές εμπορίας, σεξουαλικού χαρακτήρα, ε, με εμπορία παιδιών ή σε σχέση με την αγορά εργασίας και μας δώσατε στατιστικά στοιχεία που μας φέρνουν σε απόγνωση ε, εμένα και πολλούς συναδέλφους γιατί είναι πολύ ε, υψηλά τα νούμερα που αναφέρατε. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποιο είναι το, ποια είναι η συνηθέστερη μορφή εμπορίας στην Ευρώπη Κατόπιν, θα μπορούσατε να μας δώσετε μία απάντηση σε σχέση με το πόσο επιτυγχάνεται η ισορροπία ανάμεσα στα μέτρα ελέγχου, ε, συνοριακού ελέγχου και των μέτρων προστασίας ε, των θυμάτων ε, εμπορίας. Δηλαδή, πώς γίνεται η διασύνδεση στην πράξη. Σας ευχαριστούμε, κύριος Μίλλερ, τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ κύριε Βασιλεύ γιατί η παρουσίασή σας ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έχω μία ερώτηση που σχετίζεται με μία συζήτηση που κάναμε σήμερα το πρωί. Ε, είπατε ότι συνεργάζεστε στενά με την ε, Frontex, ε, με τη Eurojust. Πολύ ωραία όλα αυτά. Υπάρχει όμως επαρκή συντονισμός. Και πιο συγκεκριμένα θα σας ρωτήσω το εξής. Κρίνετε ότι ενδείκνεται να διοριστεί ένας ε, εισαγγελέα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αναλάβει ακριβώς αυτό το συντονιστικό ρόλο των επιμέρους οργανισμών. Η ε, κυρία Μορβάη τώρα. Σας ευχαριστώ Ζητώ συγγνώμη ε, που δεν άκουσα την προφορική σας ε, παρουσίαση γιατί είχα λυμμένες υποχρεώσεις. Είχα όμως ε, το προνόμιο να συσκεφτώ μαζί σας πρόσφατα και διάβασα αυτό το σημαντικό έγγραφο για τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων οι Ούγγροι και άλλοι που ζουν στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλό θα ήταν να διαβάσουν αυτή την έκθεση διότι υπάρχουν μεγάλες οικονομικές ανισότητες και ως εκ τούτου ε, ανήκουν σε επαθείς ομάδες και αναγκάζονται να μετικήσουν, να εγκαταλείψουν τις οικογένειές τους και να εξερευνήσουν ποιες δυνατότητες απασχόληση υπάρχουν σε άλλα κράτη-μέλη, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αρκετά συχνά είναι πολιτικά λεπτό αυτό το ζήτημα. Σπάνια αναφέρεται αυτό. Όταν μιλάμε για την εμπορία ανθρώπων, ε, για την αγορά εργασίας, ε, είναι δύο ε, τα βασικά ζητήματα Εφενός έχουμε ανθρώπους από τρίτες χώρες, από τον, σε εισαγωγικά τρίτο κόσμο που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέφτουν θύματα εμπορίας και ε, ε, τους εκμεταλλεύονται, υπάρχουν καταχρήσεις, είναι μια μοντέρνα σκλαβιά. Και από την άλλη έχουμε δευτεροκλασάτες χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την περιφέρεια κυρίως της Ένωσης, όπως και η δική μου χώρα, η Ουγγαρία, ε, πρώην ε, σοσιαλιστικές ε, χώρες και άλλες χώρες στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περιέλθει σε μια κατάσταση που είναι παρεμφερής με αυτή του τρίτου κόσμου ενώ υποτίθεται ότι είμαστε ισότιμοι εταίροι στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολίτες των χωρών μας ε, λόγω των συνθήκων αναγκάζονται να μετικήσουν και να ε, εξερευνήσουν δυνατότητες απασχόλησης σε πλουσιότερες, φορότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. το συνολικότερο πλαίσιο τίθεται ως ε, αυτό της μετανάστευσης. Το δεύτερο όμως οι Ανατολικοευρωπαίοι που μετικούν στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκής Ένωση ε, για καλύτερε δυνατότητε απασχόλησης. Εκεί τίθεται ένα διαφορετικό πλαίσιο ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Δεν πρόκειται πλέον για μετανάστευση. Ε, η μη κατοχήρωση των δικαιωμάτων τους, ε, η ευπαθής του θέση και η καταπίεση αυτών των ανθρώπων αναγνωρίζεται σε πολύ μικρότερο βαθμό ε, σε σχέση με όσους θεωρούνται μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πρεσβεύετε εσείς γι' αυτό και κατά τη γνώμη σας πώς θα μπορούσαμε να φέρουμε κάποιες αλλαγές σε αυτή την δινή κατάσταση συχνά, Ούγγροι, έρχονται σε επαφή με μένα διότι προσπαθούν ε, να βρουν μια θέση απασχόληση ε, σε χώρες Δυτικής Ευρώπης, ε, εργάζονται σε συνθήκες δουλείας, δεν αμείβονται σωστά, εργάζονται σε χείριστες συνθήκες και έχουν ακόμη μικρότερη θεσμική νομική προστασία σε σχέση με μετανάστες από τρίτες χώρες δεν έχουν ε, ε, ε, κυβερνητικά όργανα ή μη κυβερνητικές οργανώσεις που να τους προσφέρουν ένα πολυσύνθετο πλαίσιο υπηρεσιών, ιατρικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες και κυρίως αλεξίου σημαντικών νομικές υπηρεσίες για να ενισχυθεί ο αγώνας τους και να προστατωθούν. Μπορεί αυτό να αλλάξει, μπορείτε εσείς να διοχετεύσετε πόρους σε αυτό αυτό το τομέα με τρόπο ώστε οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύονται και να αναγνωριστεί και αυτό το πρόβλημα, να αναγνωριστεί η σοβαρότητά του. Ποιο... θα ήταν το μήνυμά σας προς τους Ούγγρους, ε, Φερρυπίν, που ε, πέφτουν θύματα Αυτέ οι εκμετάλλευση και στερούνται δικαιωμάτων και δεν ε, έχουν νομική προστασία που προσφέρεται σε πλουσιότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερμανία. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα τώρα. Μία συγκεκριμένη περίπτωση στην Ισπανία, μια συγκεκριμενη περιπτωση στην ισπανια μια ογκαρέζα, ε, η οποία ε, προσπαθούσε να βρει δουλειά έπεσε θύμα εμπορίας και την εκμεταλλεύτηκαν βάναυσα, οι Ισπανικές αρχές ε, τη βοήθησαν, άρχισε η ποινική δίωξη στην Ισπανία και εκείνη επέστρεψε στην Ουγγαρία. Όμως οι Ουγγρικές αρχές αυτή τη στιγμή λένε ε, ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτή τη γυναίκα διότι έπεσε θύμα εμπορία στην Ισπανία και ως εκ τούτου οι Ισπανικές αρχές είναι αυτές που είναι αρμόδιες. Λοιπόν, ε, τώρα δεν δικαιούται ε, ιατρική ασφάλιση, ψυχολογική υποστήριξη, ε, αποζημίωση, διότι οι ισπανικές ε, αρχές δεν τις προσέφεραν αποζημίωση, δεν την ενημέρωσαν για το δικαίωμα προς αποζημίωση και τις είπανε τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Σύντομη ερώτηση λοιπόν ο βασικός ε, λόγος για την σεξουαλική εκμετάλλευση πιστεύετε ότι είναι το φαινόμενο της πορνείας, ότι αν δεν υπήρχε πορνεία δεν θα υπήρχε και εμπορία για λόγους σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ε, είστε σε επαφή με το λόμπι των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν στόχο να πάψει το φαινόμενο της πορνείας και ότι θα έπρεπε να στοχεύουμε και τα δύο ταυτόχρονα καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων για λόγους σεξουαλικής εκμετάλλευσης και καταπολέμηση της ίδιας της πορνείας. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Βασιλιάδου, είναι μεγάλη πίεση γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Ε, και έχουμε και προγραμματισμένο χρόνο για τη συζήτηση, δεν μπορούμε να τον υπερβούμε. Δεν μπορείτε να επισέλθετε σε λεπτομέρειες ε, για όλα τα επιμέρους ερωτήματα. Βάλτε τα δυνατά σας και προσπαθήστε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις μπορείτε, στο μέτρο που μπορείτε. again. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η γνώση και το ενδιαφέρον αυτού του Κοινοβουλίου από όλε τι πολιτικέ οικογένειε και αυτό έχει θεμελιώδη σημασία. Θα προσπαθήσω να απαντήσω κάποιε από τι ερωτήσει. Πρώτον, όσο αφορά τα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την περίοδο 2008, 9 και 10. Όλο και περισσότερο τα στοιχεία που λαμβάνουμε βελτιώνονται. Η ποιότητά τους είναι καλύτερη σε τομείς που τα κράτη-μέλη μπορούν να ανταποκριθούν. Ε, περνούμε και εμείς λοιπόν, αλλά και τα κράτη-μέλη, μια διαδικασία μάθησης και τα κράτη-μέλη πρέπει να εξοικειωθούν. Ε, τώρα για την Ισπανία, το μόνο που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Όσο αφορά την αύξηση του αριθμού, υπάρχουν δύο εξηγήσεις. Η μία είναι να εντείνεται το φαινόμενο, γιατί μερικές φορές ε, τα φαινόμενα αυτά έρχονται σε κύματα και η οικονομική κρίση τα επιδεινώνει ή μπορεί οι ισπανικές αρχές να βελτιώθηκαν στην ε, εξακρίβωση των θυμάτων και των δικτύων ή μπορεί να συνεπάρχουν οι δύο παράγοντες. Όσο αφορά τις καταδίκες, πραγματικά είναι ένας στόχο στον οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε κατά την ελοποίηση της οδηγίας. Γιατί η μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών είναι ένα πράγμα, αλλά μετά η υλοποίηση της οδηγίας είναι ένα άλλο θέμα. Θα πρέπει να δοθεί βοήθεια και διευκόλυνση στις αρχές των κρατών μελών, να διευκολυνθεί η δίωξη και η καταδίκη. Και φυσικά χρειάζεται πολλές φορές διακρατική ε, συνδρομή, για παράδειγμα με τις χώρες προέλευσης. Είναι κάτι που μπορεί να επιδιωχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε σχέση με τη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, όπως σας είπα, εννέα κράτη-μέλη ειδοποίησαν ε, μερικοί Ε, μεταφορά της οδηγίας. Τα κράτη-μέλη έχουν ενημερωθεί ε, και υπάρχει και έλλειψη επικοινωνίας με 13 κράτη-μέλη. Φυσικά θέλουμε να διασφαλίσουμε την ορθή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και θα ξεκινήσει και διαδικασία επί του κοινοτικού δικαίου κατά των κρατών μελών εάν δεν την ε, ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο. Σίγουρα εσείς είστε πιο ενήμεροι από εμένα πάνω σε αυτό, αλλά το Κοινοβούλιο έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον και πολιτική βούληση για το θέμα αυτό. Και πραγματικά έχει έρθει η ώρα να κάνουμε και περισσότερα, οπότε ίσως να γίνουν τέτοιες διαδικασίες. Τώρα, για τα παιδιά και μονομένους τομείς όπου δραστηριοποιούμεθα, ε, όχι μόνο δίνουμε πολύ μεγα... εξετάζουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το θέμα των παιδιών, ε, και δεν εστιαζόμαστε μόνο στο τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στο τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη καλούνται να στήσουν προστατευτικές δομές για τα παιδιά. Στις επόμενες μέρες θα δημοσιευθεί ε, μία πρόταση για την αντιμετώπιση της επαιτίας, ε, της καταναγκαστικής επαιτίας. Όχι μόνο είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό, αλλά είναι και ένα θέμα που πρέπει να το εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Ε, η μελέτη διαπίστωσε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στον ορισμό, στους ορισμούς που υπάρχουν. Αυτό πριν από τη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη σαφήνεια στους ορισμούς. Όσο αφορά τις πληθυσμούς Ρωμά, ε, συμμετέχουμε ε, πάρα πολύ ε, στο έργο των συναδέλφων από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης για τους Ρωμά Υπάρχει όχι μόνο μία, αλλά τουλάχιστον μία οργάνωση γυναικών Ρωμά που εργάζεται άμεσα και ειδικά με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και θα έρθουν στην πλατφόρμα την Παρασκευή. Ήρθαν στην πλατφόρμα την Παρασκευή. Ε, θα κάνουμε μια μελέτη για τις ευάλωτες ομάδες και φυσικά οι Ρωμά και ιδίω τα παιδιά θα έχουν ε, την πρωτοκαθεδρία εκεί. Γιατί προφανώς ε, υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό καταναγκαστικής εποπτείας μεταξύ των πληθυσμών αυτών. Όσο αφορά το έργο των ακαδημαϊκών, Νομίζω ότι το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε ξεκινήσει μια μελέτη με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας προϋπολογισμού 2.500 ευρώ, 2,5 ε, εκατομμυρίων ευρώ και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη γενική διεύθυνση για να γίνει αυτό. Γιατί πραγματικά πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ρίζες, πού ερίζεται η ζήτηση για την εμπορία των ανθρωπίνων όντων και ποια είναι η καλύτερη πολιτική αντιμετώπισης των προβλημάτων. Ε, εμένα, ε, εγώ υπήρξα ακαδημαϊκός ε, επί 15 χρόνια και φυσικά και το έργο των ακαδημαϊκών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε σχέση με την προστασία της εργασίας και τους επιθεωρητές εργασίας υπάρχει ένα παραδοτέω με την Eurofound, άλλον ευρωπαϊκό φορέα, τον 8ο με τον οποίο συνεργαζόμαστε και πολύ στενά μάλιστα. Αυτό που θέλω να δω στην εκμετάλλευση της εργασίας και ελπίζω ότι απαντώ σε περισσότερες, τις μη, περισσότερες ερωτήσεις. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε καλύτερα ε, Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές ε, για, την, ε, για τον τρόπο που εργάζονται επιθεωρητές εργασίας, αλλά και πώς ε, εφαρμόζονται τα εργασιακά δικαιώματα στο κάθε κράτος μέλος. Καταρχήν πρέπει το κάθε άτομο να είναι ενήμερο για τα εργασιακά του δικαιώματα για να μπορέσει να τα διεκδικήσει. Είναι η αφετηρία αυτό. Τώρα, Όσο αφορά ε, τις χώρες δεύτερης κατηγορίας, όπως εσείς τις αποκαλέσατε, το 61% των θυμάτων, και μιλάω για στοιχεία που μας έχουν δώσει επισήμως τα κράτη-μέλη, ε, είναι εσωτερικά θύματα, δηλαδή θύματα που είναι Ευρωπαίοι πολίτες και επειδή διακινούνται παράνομα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποθέτω ότι η συζήτηση για το κατά πόσο τα θύματα είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνεται διάκριση. Πρέπει και δύο κατηγορίες ε, να αντιμετωπίζονται. Τώρα το θέμα του grooming, της προσέγγισης νεαρών κοριτσιών μέσω της ε, το ότι δήθεν ε, οι προαγωγοί ερωτεύονται τις κοπέλες αυτές. Ε, παρακολουθώ τα δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου. Ε, φυσικά είναι παράνομη αυτή, αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς και φυσικά πρέπει να γίνει κάτι. Τώρα αυτό που λέτε η συνιστόσα της μεταφοράς ατόμος, ατόμων για να υπάρχει το αδίκημα της ε, εμπορίας ανθρωπίνων όντων, πάντοτε υπάρχει κάποιος τύπου μεταφοράς έστω και στο εσωτερικό των κρατών μελών. Φυσικά πρέπει να τα συζητήσουμε περισσότερο αυτά δεν έχω απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Τώρα για την παροχή βοήθειας προς τα θύματα. Υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις και στη στρατηγική και στην οδηγία. Δεν λέω ότι αυτό είναι η αρχή και το τέλος, ότι όλα αρχίζουν και όλα τελειώνουν εκεί. Αλλά νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ καλό θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο. Εκείνο που δεν είναι καλό είναι η υλοποίηση και η εφαρμογή τους. Και ακριβώς εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, στην καλύτερη υλοποίηση όλων των άρθρων της οδηγίας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις για την παροχή βοήθειας. Τούτου λεχθέντος πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πολλοί από τους ανθρώπους που διακινούνται παράνομα και διασώζονται, ξαναεπιστρέφουν στην παράνομη διακίνηση ανθρωπίνων όντων μετά. Τώρα, σεξουαλική κακοποίηση και πορνεία και η σχέση τους. Είναι σαφέστατη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια έντονη θητεία να δράσεις όσο αφορά για την, την εμπορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν έχει θητεία για την... Δεν έχει εντολή να δράσει στον τομέα της πορνείας. Ε, φυσικά τα δύο συνδέονται. Όταν η, η πορνεία ε, συνεπάγεται την εμπορία ανθρωπίνων όντων, τότε ναι, εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την αρμοδιότητα να ε, επέμβει. Ε, πριν από μερικές, μερικούς μήνες ε, ήμουν εδώ σε μια διάσκεψη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θυμάμαι ότι υπήρχαν 200 οργανώσεις της ε, τοπικής κοινωνίας που είχαν συμμετέχει Υπάρχουν πολλές ιδεολογίες βέβαια και θέλουμε οργανώσεις από όλο το φάσμα της κοινωνίας των πολιτών για να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο ε, με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά στο κάθε κράτος μέλος. Φυσικά δεν είμαστε αρμόδιοι να μιλήσουμε για την πορνεία. Υπάρχει κρίκος μεταξύ εμπορίας και πορνείας και τον εξετάζουμε προσεκτικά. Ζητώ συγγνώμη που δεν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, με χαρά μου να να απαντήσω εγγράφω ή ηλεκτρονικά σε άλλες ερωτήσει που τυχόν μου αποστείλετε αργότερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ε, ζητούμε συγγνώμη που επισπεύδουμε έτσι την, ε, το κλείσιμο της συζήτηση, Έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Προσπαθήσατε να απαντήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ερωτήσεις μέσα στον χρόνο. Ε, υπερβήκαμε τα χρονικά μας όρια και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο ε, θέμα. Θα παρακολουθούμε όμως τις επιδόσεις της υπηρεσίες σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ready to go. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να συνεχίσουμε. Το επόμενο σημείο, το σημείο 10. Εφαρμογή της στρατηγικής για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμουν εγώ εισηγητής για το θέμα αυτό για να παρουσιάσω το σχέδιο ψηφίσματος για τη δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή αυτή τη ε, στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συντονιστέ ε, αποφάσισαν να λάβουν θέση αντιδρώντα τη δεύτερη έκθεση για την εφαρμογή τη στρατηγική που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο με μια προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια. Και στη συνέχεια θα ακολουθούσε μια συζήτηση που θα κατέληγε σε ένα ψήφισμα που θα το προετοίμαζε η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Και σήμερα εδώ συζητάμε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια σύντομη εισαγωγή αυτού του σχεδίου ψηφίσματος. Βασίζεται καταρχήν στην έκθεση της συναδέλφου κυρίας Μπορσελίνο που συντάχθηκε πέρυσι για, την εσωτερική, για τη στρατηγική εσωτερική ασφάλειας και αναπτύσσει τα σημεία της έκθεσης Μπορσελίνο Καταρχήν, συμπεριλαμβάνει κάποιες σκέψεις για τον κύκλο πολιτικής και τις πιθανές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Δεύτερον, ε, περιλαμβάνει κάποια συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν στην ε, διάμεση έκθεση ΚΡΙΜ και μια πρώτη αντίδραση ε, στην έκθεση της ΟΚΤΑ για το σοβαρό οργανωμένο έγκλημα και την έκθεση για την κατάσταση της τρομοκρατίας και τις σχετικές τάσεις, την έκθεση ΤΕΣΑΤ που παρουσιάστηκε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πρόσφατα διαμορφωμένη η έκθεση αυτή από τη Europol. Καθώς επίσης και κάποιες ιδέες για τη συνέχιση που θα δοθεί στην ε, στρατηγική εσωτερική ασφάλειας μετά το 2014 και για τον ρόλο του Κοινοβουλίου στον προσδιορισμό αυτής της νέας στρατηγικής. Έχουμε περίπου μισή ώρα για τη συζήτηση και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε σχόλια, θέσεις, παρατηρήσεις από βουλευτές ή από την Επιτροπή ή από την Προεδρία του Συμβουλίου, εάν κάποιος εκπροσωπεί την Ιρλανδική Προεδρία. Δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια. Κανείς δεν θέλει το λόγο. Κυρία Ματία, σας ευχαριστώ που έρχεστε να με βοηθήσετε σε αυτή την απόγνωση στην οποία βρίσκομαι λήψη ομιλητών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να υποκινήσουν το ενδιαφέρον και άλλων και να λάβουν και άλλοι το λόγο γιατί είναι ένα ιδιαίτερα λεπτό θέμα. Και εξάλλου σας ευχαριστώ που ασχοληθήκατε εσείς με το θέμα ως εισηγητής. Ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε για το ψήφισμα αυτό. Πολλές είναι οι ιδέες σε αυτή την πρόταση ψηφίσματος. Το είχαμε αναφέρει στις συνεδρίες των συντονιστών όπως είπατε. Είναι πολλά τα σημεία που προέρχονται και από την έκθεση Μπορσαλίνου αλλά και από την έκθεση Σόκτα που είναι πολύ σημαντική και που μας είχε παρουσιαστεί στην Επιτροπή για την εσωτερική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη βελτίωσή της. Είναι ρόλος μας στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να προχωρήσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Οι παρατηρήσει που γίνονται στο ψήφισμα για το οργανωμένο έγκλημα, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι εύστοχε. Ε, και άλλο ένα θέμα είναι το ξέπλυμα χρήματος, γιατί και αυτό συνδέεται άμεσα με το οργανωμένο έγκλημα. Και κάποιοι συνάδελφοι είναι και μέλη της Επιτροπής Κρίμου, όπως υπενθυμίσατε. Υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το συζητήσαμε, συζητήσαμε την ριζοσπαστικοποίηση των νέων, που είναι πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να το επισημάνουμε στο ψήφισμα αυτό. Να αναφέρουμε και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ώστε να ανοιχνεύεται καλύτερα η τρομοκρατία και να αποτρέπεται. Ακόμη πρέπει να τονίσουμε το βασικό ρόλο που παίζουν οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Η Europol, η Eurojust, η CEPOL και είναι πολλά τα τρέχοντα θέματα για την ανεξαρτησία αυτών των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθούν να εξασφαλίσουν καλύτερη εσωτερική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί γνωρίζουμε ότι η παραποίηση των τσιγάρων και το λαθρεμπόριο τσιγάρων είναι ο τομέας ε, με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στην παραποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσαμε να έχουμε σημαντικά φορολογικά έσοδα. Θα μπορούσαμε να λάβουμε μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθεί το λαθρεμπόριο τσιγάρων και η παραποίησή τους. Στην Επιτροπή ΚΡΙΜ είχα οργανώσει μια ακρόαση για την ε, εμπορία πυροβόλων όπλων ε, και ξέρετε ότι είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Europol και τα κράτη-μέλη, τουλάχιστον έτσι μας είπε ο εμπειρογνώμων της Europol, ότι τα κράτη-μέλη δεν είχαν πολλά δεδομένα όσον αφορά τα όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται σε δολοφονίες παραδείγματος χάρη, ε, όπως οι δολοφονίες που ξέρουμε στη Γαλλία, στη Μασαλία ή στην Κορσική, αλλά και σε άλλες χώρες υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα. Σίγουρα από κάποια σύνορα περνάνε κάποια όπλα, καλάσνικοφ και άλλα, αλλά δεν ξέρουμε πού προέρχονται τα υπόλοιπα πυροβόλα όπλα και η Europol μας είπε ότι τα κράτη-μέλη δεν τους δίδουν τέτοια δεδομένα. Θα μπορούσαμε λοιπόν επί τη ευκαιρία αυτού του ψηφίσματος να ζητήσουμε να δίνουν τα κράτη-μέλη τέτοια στοιχεία, να συγκεντρώνουν καταρχήν τέτοια στοιχεία και να, μετα... να τα μεταβιβάζουν στη Europol, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την... το θέμα της εξέτασης της εμπορίας όπλων. Αυτά κύριε Πρόεδρε και ελπίζω η δική μου παρέμβαση να παρακινήσει και άλλους να λάβουν το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος σημειώνουμε τις παρατηρήσεις σας, ιδίως αυτό το οποίο είπατε για την εμπορία όπλων. Θα δούμε τι προφυλάξεις πρέπει να ληφθούν σε αυτό το θέμα. Έχουμε μοιράσει το σχέδιο ψηφίσματος. Και αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, να σας αναγγείλω την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 3η 4 η Ιουνίου, 12 η ώρα το μεσημέρι. Ψηφοφορία στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ προβλέπεται για τις 19 ή 20 Ιουνίου. και προβλέπεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ιουλίου και να ψηφιστεί εκεί στην Ολομέλεια. Ας περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα της εφαρμογής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφαρμογή της απόφασης ΠΡΟΥΜ και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Ανταλλαγή Πληροφοριών. Έχουμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση. Έχουμε ένα ε, δεύτερο σχέδιο ψηφίσματος ε, για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας. Είναι η εφαρμογή της απόφασης Πρύμ, όπως είναι γνωστή, που είναι ένα σημαντικό ορόσημο για τη δημιουργία του χώρου δικαιοσύνης και ασφάλειας που ξεκίνησε από τη συνεργασία των κρατών μελών για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και η Επιτροπή υπέβαλε τις απόψεις της πέρυσι το Δεκέμβριο. Οι συντονιστές για το θέμα αυτό αποφάσισαν να υποβληθεί ένα προφορικό ερώτημα και να γίνει μια συζήτηση στην Ολομέλεια που θα καταλήξει σε ένα ψήφισμα το οποίο θα προετοιμάσει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Το σχέδιο ψηφίσματος λοιπόν περιλαμβάνει πρώτον την τωρινή κατάσταση των διαφόρων οργάνων, διάβλων και εργαλείων για ε, την ε, ενημέρωση σχετικά με την επιβολή του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνοριακό επίπεδο και λέγεται ότι είναι πολύπλοκο αυτό το τωρινό τοπίο και αυτό οδηγεί σε αναποτελεσματικότητες ε, και ανεπαρκή δημοκρατική εποπτεία. Δεν είναι λοιπόν ικανοποιητική η κατάσταση και ε, έχουν ακουστεί πολλές ε, επικρίσεις. Δεύτερον, η Επιτροπή κατέγραψε την τρέχουσα κατάσταση. Φαίνεται ότι έχουν χαθεί πολλές ευκαιρίες Άρα μας χρειάζεται ένα μελλοντοστραφές όραμα, πιο φιλόδοξο, για το πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε ε, την κοινή χρήση δεδομένων για την επιβολή του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγγυόμενοι ένα ε, καλό επίπεδο προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας, κάτι το οποίο ζητούσε και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, και η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Τρίτο σημείο που περιλαμβάνεται είναι ότι ε, πολλά από τα μέσα αστυνομικής συνεργασίας εγκρίθηκαν υπό τον τρίτο πυλώνα, τον πρώην τρίτο πυλώνα. Παράδειγμα είναι η απόφαση Προύμ. Αλλά ακόμη δεν υπάρχει η σωστή δημοκρατική εποπτεία και έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη θέσπιση της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να έχει αυτόν τον έλεγχο. Πρέπει λοιπόν αυτά τα μέσα να ευθυγραμμιστούν με το νομικό πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας και η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις σύντομα, ούτω ώστε αυτά τα όργανα του πρώην τρίτου πυλώνα να ακολουθήσουν την τωρινή στρατηγική στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτή είναι η κατάσταση και τώρα θα συζητήσουμε ακριβώς αυτό το σχέδιο ψηφίσματος. Θέλει κανείς το λόγο? Υπάρχουν σχόλια? Δεν υπάρχουν σχόλια. Σήμερα το απόγευμα φαίνεται ότι είμαστε τυχεροί. Δεν ξέρω γιατί. Εν δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια. Έχει διανεμηθεί το ψήφισμα σε όλες τις ομάδες και σε όλους τους βουλευτές. Αν δεν υπάρχουν σχόλια και δεν έχει ούτε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής κάποιο σχόλιο, περνάμε στην προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Θέλει κάτι να πει η Επιτροπή, όχι. Λοιπόν, προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών είναι 3η 4 Ιουνίου, 12 το μεσημέρι ώστε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών 19 με 20 Ιουνίου και να πάει στην Ολομέλεια του Ιουλίου. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλα σχόλια, οπότε ολοκληρώθηκε και αυτό το θέμα. Και περνάμε στο σημείο 12, ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος της Στοκχόλμης. Εδώ έχουμε συνεργασία τριών επιτροπών που είχαν ασχοληθεί αρχικά όταν πρώτο συζητήσαμε το θέμα και καταλήξαμε στην υιοθέτηση του αποκαλούμενου προγράμματος της Στοκχόλμης και δόθηκε εντολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο του 2009 επί Σουηδικής Προεδρίας. Υιοθετήθηκε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, ήταν το τρίτο κεφάλαιο αυτής ε, της συνεχιζόμενης τριτού στρατηγικής για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Τώρα αυτό είναι πλέον ευρωπαϊκή πολιτική και θα πρέπει να ακολουθήσει την νομοθετική διαδικασία της συνθήκης της Λισαβόνας και οι τρεις επιτροπές που είχαν ασχοληθεί αρχικά, η Συνταγματική Επιτροπή, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, τώρα θα ασχοληθούν με την ενδιάμεση αξιολόγηση αυτού του προγράμματος. Κάπως καθυστερημένα, όπως θα παρατηρήσετε γιατί έχουμε ήδη περάσει το σημείο της ενδιάμεσης ε, αξιολόγησης. Ένας χρόνος έχει μείνει, έχουμε φτάσει στο τέλος αυτού του διαστήματος, αλλά εν πάση ακόμη έχουμε χρόνο να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Να δούμε πώς απέδωσαν αυτά τα οποία θεσπίστηκαν κατά τα περασμένα τέσσερα χρόνια. και να δούμε τι διδάγματα υπάρχουν και τι συμπεράσματα μπορούμε να εξαγάγουμε. Λοιπόν, μια συνεργασία των Επιτροπών ΑΦΚΟ, Γιούρι και ΛΥΜΠΕ σύμφωνα με τον ε, κανονισμό Θα αντιμετωπίσουν λοιπόν αυτές οι τρεις επιτροπές από κοινού το έργο της ενδιάμεσης αξιολόγησης. Οπότε εδώ ο ρόλος μας είναι η ανταλλαγή απόψεων και αποφασίσαμε να συζητηθεί το έγγραφο εργασίας και εγώ ως πρόεδρος ανέλαβα να είμαι εισηγητής αυτού του θέματος και γι' αυτό σας το υποβάλλω προς συζήτηση. Να σας υπενθυμίσω τις βασικές ιδέες. Καταρχήν, εδώ θέλουμε να κάνουμε μία συζήτηση, τίποτα παραπάνω. Κάναμε μία πρώτη συζήτηση με τους κοιόδης συζήτητες. Συμφωνήθηκε καταρχήν η βασική προσέγγιση με τους συνεισηγητές από τη Γιούρη ο κύριος Μπελιγκουέρη και από την ΑΦΚΟ ο κύριος Καρλοκαζίνη. θα ξεκινήσουν τις συζητήσεις και στις αντίστοιχες επιτροπές και με βάση τις συζητήσεις αυτές θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης. Θέλουμε να αξιολογήσουμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, όπως σας είπα. να αποκομίσουμε μια συνολική εικόνα, διότι αυτό είναι κάτι που δεν το κάνουμε πολύ συχνά. Να δούμε το χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας με ένα ολιστικό τρόπο, ξεκινώντας από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. για να συζητήσουμε τουλάχιστον τρία πράγματα στη διαδικασία αυτή. Πρώτον, να δούμε αν όντως έχουμε δώσει κάτι απτό στους πολίτες, γιατί μιλάμε για δικαιώματα, μιλάμε για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, μιλάμε για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το Σέγγεν, για το άσυλο, αστυνομία, αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Έχουμε δώσει κάποια αυτά αποτελέσματα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, το 2013 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών. Ένα θέμα που μας αφορά όλους. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μία δημόσια συζήτηση, να προάγουμε μία συζήτηση σε ολόκληρη την Ευρώπη και να εμπλακούν και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. ώστε να συγκεντρώσουμε τα σχόλια της κοινωνίας των πολιτών για τα αποτελέσματα του προγράμματος της Στοκχόλμης κατά τη γνώμη τους και για τις πιθανές βελτιώσεις του περιεχομένου του προγράμματος στο μέλλον. Και το τρίτο σημείο είναι το αν θα πρέπει να υπάρξει και διάδοχος του προγράμματος της Στοκχόλμης. Το 1999 είχαμε το Τάμπερ, θυμάστε, μετά είχαμε τη Χάγη, το 2004. Τώρα έχουμε τη Στοκχόλμη. Για πέντε χρόνια. Βέβαια το πρόγραμμα της Στοχόλμης ε, θεωρήθηκε ότι θα είναι ένα ορόσημο. Γιατί εδώ είχαμε ενισχυμένη συνεργασία σε θέματα που ήταν θέματα κυριαρχίας των κρατών μελών πιο πριν. Μετά την συνθήκη της Λισαβόνας είναι ευρωπαϊκά αυτά τα ζητήματα και δεν θέλουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν, αλλά έχουμε εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο να κάνουμε πράγματα, να συνεργαστούν η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να λαμβάνουν πρωτοβουλίες. Να δεσμευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει συγκεκριμένα βήματα προς τους στόχους της συνθήκης της Λισαβόνας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα διάδοχο του προγράμματος της Στοκχόλμης. Αυτό είναι ένα θέμα για ανοιχτή συζήτηση. Κάτι που το συζητήσαμε στο Στρασβούργο και η Ιρλανδική Προεδρία τόνισε τη σημασία του πολιετούς προγράμματος για να διασφαλίσουμε τη συνοχή και συνεκτικότητα την χάραξη πολιτικών από τις ε, προεδρίες της Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θέλουμε να έχουμε ένα πρόγραμμα που θα δίνει πολιτική όθηση και δυναμισμό και ταυτόχρονα είναι καθήκον μας να συνεργαστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Προσπαθήσαμε, αλλά δεν τα πολύ καταφέραμε μέχρι τώρα. Άρα υπάρχουν σημεία προς συζήτηση που θα πρέπει ανοιχτά να τα συζητήσουμε για να είναι και χρήσιμα. Λοιπόν, θέλουμε μια στρατηγική για μετά τη Στοκχόλμη. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα είναι αυτή η στρατηγική. Δεν ξέρουμε πώ μπορούμε να την εξειδικεύσουμε αυτή τη στρατηγική, Πάντω χρειαζόμαστε μια στρατηγική. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο και αυτό είναι σίγουρο. Και η μόνη πιθανή πορεία είναι να ακολουθήσουμε το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είχε διαμορφωθεί βάσει της παλιάς συνθήκης, βάσει του παλαιού θεσμικού πλαισίου. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στο μέλλον. και με νέες ιδέες τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν κάποιο ρόλο για αυτό το χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε πριν συντάξουμε την πρώτη έκθεση ως αποτέλεσμα της ζητήσεως που θα κάνουμε, όπως σας είπα, σε συνεργασία, εγώ και οι συγητές από την Επιτροπή Γιούρη και ΑΦΚΟ, μετά από αυτόν τον πρώτο γύρο συζητήσεων. Και τώρα έχετε εσείς το λόγο για να υποβάλλετε παρατηρήσεις και σας παρακαλώ να υποβάλλετε παρατηρήσεις για να με βοηθήσετε στη δουλειά που έχω να κάνω. Βλέπω κάποιον που ζητά το λόγο. Ευτυχώς, εδώ κάποιος θέλει το λόγο. Με σώσατε γιατί τα προηγούμενα θέματα σήμερα το απόγευμα δεν υποκίνησαν μεγάλη συζήτηση. Ο κύριος Μπρόνς και μετά η κυρία Μόρβαη. I'm sorry, I'm sorry. I No, I'm sorry. If you allow me... Ζητώ συγγνώμη. Ε, ο κύριος Κίρκοπ είχε ζητήσει πρώτος το λόγο, αλλά εγώ δεν τον είχα δει. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Μπρόνς. Ε, συγγνώμη, πρόεδρε. Δεν ήθελα να διαταράξω τη συζήτηση, ήθελα μόνο να αντιδράσω σε σχέση με τα σχόλια που κάνατε γενικότερα για το πρόγραμμα της Στοκχόλμη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία πως ε, παρότι θα υποστήριζα τα, όλα τα επιμέρους στοιχεία του προγράμματος, ε, είναι σημαντικό να έχουμε και ένα θεματολόγιο, ένα προγραμματισμό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατεύσουμε και τις μεθορίους μας και τους πολίτες μας. Στη στρατηγική Στοχόλμη υπάρχουν διάφορα σημεία που ε, τελικά είχαν ε, θετικά, αρκετά θετικά αποτελέσματα. Η στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια πρώτα απ' όλα. Ε, πέραν κάθε αμφιβολία, είδαμε ξεκάθαρα σημάδια πρακτική συνεργασία ανάμεσα στι αρχέ επιβολή του νόμου ε, κατά τις οργανωμένες εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας κυρίως ζήτησαν ε, δράση κατά της ε, κατάχρησης των δικαιωμάτων ελεύθερης μετακίνησης από πολίτες τρίτων χωρών και αυτό είναι θετικό. Θα έπρεπε επίσης να καλωσορίσουμε νομίζω την γενική προσέγγιση για τα θέματα ασύλου από νομοπαρασκευαστική πλευρά, γιατί προστασία των δεδομένων, γιατί το πρόγραμμα Στοχόλμης ε, έτσι άρχισε. Θέλαμε να βρούμε μια εξορυπμένη προσέγγιση και στον τομέα του ασύλου. Είναι προφανές και νομίζω αναμενόμενο ο μου ότι ε, δηλώνω απογοητευμένος για τα ζητήματα ε, του PNR, δικαιώματα και στοιχεία επιβατών, καθώς και για ζητήματα δημοσίου τάξης. Ελπίζω ότι θα είχαμε σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο μέχρι στιγμής. Όμως ε, ε, είπατε ότι καλό θα ήταν να εξετάσουμε τα μελλοντικά μας βήματα. Λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό του προγράμματος του Στοχολ, της Στοχόλμης ε, ήταν η εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας για όλες τις δράσεις. Είναι σημαντικό όμως να μην παραφορτώσουμε και το πρόγραμμα και μην ξεχνάμε ότι στην ε, τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία έχουμε ε, κρεμούν πολλά πράγματα ακόμη. Άρα θα πρότεινα να το έχουμε όλοι κατά νου και να προβληματιστούμε για τις επιτυχίες που έχουν σημειωθεί, τις οποίες ανέφερα και εγώ και σίγουρα θα το κάνουν και άλλοι όμως, στο σημείο που φτάσαμε, ας επανεστιάσουμε τις προσπάθειές μας σε κάποιες ε, βασικές πρωτοβουλίες που δεν έχουμε φέρει σε πέρας. Ή να αναθεωρήσουμε, ε, να εξετάσουμε σε ποια σημεία υπολείπεται σοβαρό έργο. Με ηρεμία όμως και χωρίς ε, να ξεχνούμε ποτέ ε, τους βασικούς μας στόχους, δηλαδή προστασία των πολιτών, όπως σας είπα στην αρχή της, προσ... της παρέμβασής μου, και προστασία των συνόρων μας. Ε, είμαι ικανοποιημένο λοιπόν με κάποια από τα στοιχεία, αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε κατά τη γνώμη μου. Σα ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο. Σα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπρόν τώρα. Σα ευχαριστούμε. Ε, πολύ ενδιαφέρον αυτό το έγγραφο εργασία. Το διάβασα και κάποια τα μάθα και απ' έξω. Όχι, αστείευομαι. Ε, στο δεύτερο τμήμα ε, μιλάτε για πιθανούς στόχους για την αξιολόγηση του προγράμματος Στοχόλμης από πλευράς Επιτροπής μας και μας ε, λέτε για την εφόσον η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ζήτημα κέρια σημασία για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και πρέπει να το δούμε από τη σκοπιά των πολιτών και μας μιλάτε για την νομικά δεσμευτική χάρτα ε, όπου ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, τίθενται στο κέντρο, στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τη σύμβαση που τώρα συλλογικά έχουμε κυρώσει, δεν έχουμε κυρώσει δηλαδή ανακράτος μέλος, αλλά έχει κυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν κάποια δικαιώματα που αντίκειται σε αυτά τα δικαιώματα της χάρτας. Προσπάθησα ε, να καταλάβω από τους εμπειρογνώμονες ακριβώς ποια είναι αυτά τα σημεία, να μου το εξηγήσουν ναι, ρητά. Ε, υπάρχουν κάποιες ελευθερίες, όλες οι ελευθερίες είναι ίσες, αλλά κάποιες είναι ισότερες, ας το πω έτσι από τις άλλες. Ε, η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης φαίνεται ότι υπερέχει σε σχέση με μια σειρά ανθρωπίνων δικαιωματών και ελευθεριών που δεν πρέπει να παραβιάζονται. Η ελευθερία για την προστασία κατά της διακριτικής μεταχείρισης φαίνεται να είναι πιο σημαντική σε σχέση με την άσκηση ε, κάποιας θρησκείας, κυρίως όταν μιλάμε για το χριστιανισμό και το είδαμε αυτό στους γάμους των ομοφιλοφίλων ε, και στο ζήτημα των οικοτροφίων. Ε, φάνηκε εκεί πέρα ότι τελικά δεν είναι ισότιμα όλα τα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε για κάποια ε, γενική αρχή επί τη βάση της οποίας ε, θα ιεραρχήσουμε τα δικαιώματα ε, διότι φαίνεται ότι υπάρχει, υπάρχουν αντιφάσεις σε ορισμένε περιπτώσεις. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπρόνς, κυρία Μορβάη. Σας ευχαριστώ. θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Κίρχοπ όταν μας λέει ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και η συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικές ε, και στις δικαστικές αρχές των κρατών μελών ε, ουσιαστικά επικεντρώνονται στο θέμα της προστασίας ε, των δικαιωμάτων των πολιτών και το 2013 είναι το έτος της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας όπως γνωρίζετε. Θα πρότεινα λοιπόν, Πρόεδρε, δεν θα έπρεπε να ρωτήσουμε και τους πολίτες για τις προσωπικές τους εμπειρίες, τα βιώματά τους κατά την εφαρμογή του προγράμματος ε, χόλμης και το πώς έχει επηρεαστεί ε, στην ουσία η καθημερινή του ζωή και κατά πόσο είναι επιτυχημένη όντως στην πράξη αυτή η συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικές και στις δικαστικές ε, αρχές. Δύο περιπτώσεις συγκεκριμένες μου που καταδεικνύουν την αποτυχία του συστήματος συνεργασίας. Θα πρέπει λοιπόν σοβαρά να σκεφτούμε το ενδεχόμενο επανεξέτασης των κανονισμών και του συνολικότερου πλαισίου. Θα έπρεπε να αποτιμήσουμε και τους λόγους αποτυχίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές. Ε, η υπόθεση Τόμπιν, ε, σας την έχω εκθέσει πολλάκις ε, και στην Ολομέλεια και εδώ στην Επιτροπή Λίμπε. Πρόκειται για έναν Ιρλανδό πολίτη που δολοφόνησε, ε, σκότωσε μάλλον ε, ε, παιδιά από την Ουγγαρία λόγω οδήγησης σε κατάσταση μέθης στην Ουγγαρία Ουγγαρία για άλλους λόγους ε, του επέτρεψε να γυρίσει στην ε, Ιρλανδία και ποτέ δεν επέστρεψε. Ε, ποτέ δεν εφαρμόστηκε η ποινή φυλάκιση ούτε στην Ουγγαρία ούτε στη χώρα προέλευση του στην Ιρλανδία. Εμεί στην Ουγγαρία αυτό που θα θέλαμε ήταν να εκτίσει την τριετή ποινή φυλάκιση είτε στην Ουγγαρία είτε στην Ιρλανδία. Όμω η Ιρλανδία αρνείται να εκτελέσει την απόφαση και τελικά δεν φέρει καμία ποινική ευθύνη. Αυτός ο άνθρωπος παρότι αφαίρεσε ε, τη ζωή δύο παιδιών 1,5 και 3 χρονών αντίστοιχα είναι μία ε, προφανής ε, περίπτωση, ε, χαρακτηριστική μάλλον περίπτωση αποτυχίας της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας. Επίτροπος Δρέντι πλάκη σε αυτή την υπόθεση και διάφοροι άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Τίποτα όμως, μηδέν στο πηλίκον. Η δεύτερη περίπτωση που επίσης φαίνεται να είναι αποτυχία της συνεργασίας ε, Ουγγαρέζα η οποία είναι παντρεμένη με έναν Γάλλο και έχουν και ένα παιδί που έχει διπλή ηθαγένεια. Υπάρχει όμως οικογενειακή βία από πόσο προκύπτει από τα στοιχεία. Ο Γάλλος ε, σύζυγος ε, αυτό που κάνει είναι ότι εξαπατά την γυναίκα και τα παιδιά για να πάνε σε κάποια εξωτικά νησιά και τους λέει είναι η τελευταία ευκαιρία για να βρούμε τη γαλήνη στο σπιτικό μας και το καθεξής και είναι στη γαλλική επικράτη, είναι υπερπόντια εδάφη και εκεί συνεχίζει και γυρίζει η γυναίκα στην Ουγγαρία και ανακαλύπτει ότι ο άντρας έχει ε, πάρει το διαβατήριό της και το διαβατήριο των παιδιών και ε, εξαναγκάζοντας την έτσι να παραμείνει ε, ξεκίνησε η διαδικασία διαζυγίου. Το αρμόδιο δικαστήριο είπε ότι το παιδί πρέπει να παραμείνει στη Μπόρα Μπόρα, νομίζω εκεί είναι πήγαν διακοπές και τι γίνεται, αυτή η γυναίκα και το παιδί είναι όμοιροι ε, σε αυτό το νησί. Πάνω από έξι μήνες ε, κρατάει αυτή η ιστορία. Έχω γράψει επιστολές ε, σε όλους τους διαθέσιμους οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τίποτα δεν συμβαίνει. Και πάλι, είναι μεγάλη αποτυχία. Ας πάρουμε ένα μεγεθυντικό φακό, ας εξετάσουμε αυτές τις περιπτώσεις και ας καταλάβουμε τι πήγε στραβά. εγώ επεξεργάζομαι τώρα αυτή την ιδέα στο μυαλό μου και για την αναθεώρηση, αναδιαμόρφωση του προγράμματος. Παρακαλώ, Πρόεδρε, να λάβετε αυτό υπόψη σας. Ε, να ακούσουμε τους πολίτες, ε, τα βιώματά τους. Ε, κάποια κράτη-μέλη θα μπορούσαν να κοινοποιήσουν δικαστικές υποθέσεις σχετικές με αυτό το ζήτημα και να μάθουμε από τα παθήματα του παρελθόντος. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Βεζιά. Ε, πρόεδρε, συγγνώμη. Έχω την εντύπωση ότι ε, μας ρωτήσατε Μα ζητήσατε να εξετάσουμε αν είναι επίκαιρο ακόμη το πρόγραμμα τη Στοχόλμη ή αν πρέπει να αρχίσουμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αναθεώρηση. Κοιτάξτε, από τη στιγμή εφαρμογή του προγράμματο, τι συνέβη είναι η θέσπιση τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Καλά, δεν είμαι και ο παδό ε, φανατική, το ξέρετε εξάλλου. Όμω ενσωματώθηκε η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων συνθήκη τη Λισαβόνα. Αυτή η χάρτα ε, είναι εφαρμοστέα για τους πολίτες Ένωσης και για όσους διαμένουν στην επικράτεια της Ένωσης. Ε, και όταν ε, διαμένουν νόμιμα, νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι τα 50 εκατομμύρια που διαμένουν παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό το ζήτημα και μου φαίνεται ότι η έκθεση Γκάλ που είναι εξαιρετική, είχα συμβάλει και εγώ, ε, ε, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αντλήσουμε συμπεράσματα σε σχέση με την ενσωμάτωση συνθήκης Λισαβόνα στις χάρτες θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ω προ το διάβημα που μα προτείνεται για την ε, αποτίμηση του προγράμματο, θα έλεγα ότι συμφωνώ σε επιτοπλίστων. Είναι προφανέ ότι οι πολίτε θα πρέπει να είναι στο κέντρο του προβληματισμού μα και ο δημόσιος διάλογος θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Δεν θα είμαι δέφανο τόσο αισιόδοξη όσο ε, η κυρία Μορβάη, γιατί στις, ε, άμα κάνουμε δημοσκόπηση δεν ξέρω αν θα ξέρουν καν ποιο είναι το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη για να αποφανθούν. Ε, ε, χρειάζεται ουσιαστικός δημοκρατικός διάλογος για αυτό το ζήτημα. Επίσης, ε, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση τρομοκρατεί τους πολίτες ε, κατά κάποιο τρόπο διότι θυμάστε εδώ στην Επιτροπή μας είχαμε εκφράσει σχετικές ανησυχίες από πλευράς Γκουε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ε, σχηματίσει μια ιδέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολιτών, αλλά έδινε την εντύπωση ότι ε, το Κοινοβούλιο δεν έχει τίποτα να πει για αυτό το ζήτημα. Και εντάξει, μας μίλησε για το Ευρωπαϊκό Έτος για αυτό το ζήτημα, αλλά καταλαβαίνετε ότι με αυτά που έχουν συμβεί ε, έχουμε αυτό το μόρφωμα μπροστά μας που δεν Ζητώ συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε διαφορετικά την Ιθαγένεια. Δεν θέλω να είμαι προκλητική, αλλά εγώ είμαι υπέρ της Ιθαγένειας ε, και της διασύνδεσής της ε, με την ε, διαμονή. 16 κράτη-μέλη αντιλαμβάνονται έτσι την Ιθαγένεια, ότι πρέπει να συνδέεται άμεσα με τη διαμονή και δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από ψευδοπροβλήματα και από φόβους. Ας περάσω τώρα στο το τρίτο τμήμα, δηλαδή ποια πρόοδος έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής. Διαβάζοντας κανείς το έγγραφό σας, ε, βλέπει όλες τις ε, λήψεις που υπάρχουν. Θα είμαι και εδώ σύντομη. Για την Ευρώπη της υπερβολικής ασφάλειας, κανένα πρόβλημα. Ε, για τα υπόλοιπα όμως ακόμη και ε, για τους στόχους ε, του προγράμματος Στοκχόλμης που είναι ένα αχνό αντίτυπο του προγράμματος ε, του Τάμπερε ακόμη και γι' αυτό υπολείπεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί σε σχέση με τις φιλοδοξίες που είχε δεδηλωμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση ναι να την κάνουμε την επαναξιολόγηση να γυρίσουμε τη σελίδα αλλά νομίζω ότι είμαστε μειοψηφία δυστυχώς Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε κυρία Βερισιά. Η Μάτιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οφείλω να σας συγχαρώ ήδη για την έκθεσή σας, η οποία, εν πάση περιπτώσει, καταγράφει τον απολογισμό όλων όσων έχουν γίνει από την αρχή του προγράμματος. Εγώ είμαι λίγο πιο αισιόδοξη από την Νικολέτ. Θεωρώ ότι δεν είναι και λίγη η πρόοδος που έχει σημειωθεί από την αρχή στο επίπεδο της ασφάλειας, της δικαιοσύνης, όσο για τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και εκεί σημειώσαμε κάποια πρόοδο. Από... Φυσικά δεν είναι καθόλου τέλεια η κατάσταση, πολλά μένουν να γίνουν ακόμη. πολλά αναμένονται ακόμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα περιμένουμε αυτό το σχέδιο για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ελπίζω να μην αργήσει. Επίσης η πρόσβαση σε δικηγόρο, οι αρμοδιότητες, η δοσηδικία. Νομίζω ότι αν υπήρχαν και αυτά, ε, τότε οι πολίτες θα είχαν ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο μπροστά τους. Ε, δηλαδή η πρόσβαση σε δικηγόρο, ε, σε υπηρεσίες δικηγόρου, σε άλλες δοσιδικίες. Κάτι έχει να πει η Επιτροπή πάνω σε αυτό, αλλά δεν έχει ακόμα πει κάτι ολοκληρωμένο. Ε, καλό θα ήταν στο Συμβούλιο να μην υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι υπάρχει μια στάση αναμονής, ότι τα πράγματα δεν κινούνται, γιατί δεν υπάρχει και προϋπολογισμός, ε, γιατί τα θέματα αυτά είναι αρκετά εμβληματικά. Ε, όπως είπατε, λέγατε κι εσείς, μήπως, είπατε κι εσείς, μήπως το Κοινοβούλιο πρέπει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Πάνε δύο χρόνια που έχει κάνει την πρόταση της η Επιτροπή ε, νομίζω ότι όντως εμείς ε, οι Ευρωβουλευτές θα πρέπει να αναλάβουμε κάποια πρωτοβουλία για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών, ε, να ανταποκριθούμε στον ρόλο μας. Για το καλό του πολίτη φυσικά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε κάποια προγράμματα για να συμπληρώσουμε αυτά που έχει κάνει η Κομισιόν. Εμένα μου άρεσε η δικαστική συνεργασία και η έμφαση που δόθηκε σε αυτό. Καλό θα ήταν να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση δικαστική στην Ευρώπη. Καλό θα ήταν. Και επίσης πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη δικαστική συνεργασία, περισσότερη προσπάθεια για την κατάρτιση των δικαστών, εσείς μιλάτε, μιλήσατε για τον πολίτη ε, και το έτος του Ευρωπαίου Πολίτη, το 2013. Η κυρία Βεγζέν έχει δίκιο. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, νομίζω ότι είναι άγνωστο στην πλειοψηφία των πολιτών. Αλλά τούτου λεχθέντος, αν μιλήσουμε στον πολίτη για όσα έχουν γίνει στον τομέα της εκπαίδευσης, της ε, διερμηνίας, της ε, δικαστικής συνεργασίας, τότε ναι, και έχουν γίνει κάποια από τα βήματα. Αν εξηγήσουμε στον κόσμο τι έχει γίνει με πολύ πιο απλά λόγια, τότε μπορεί να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο. Να καταλάβουν οι πολίτες ότι η Ευρώπη είναι πολύ περισσότερο στο πλευρό τους μέσα στην καθημερινότητά τους. Απλά πρέπει να το κάνουμε αυτό με μια απλή προσέγγιση, με απλά λόγια. Δεν είμαι λοιπόν τόσο απεσιόδοξη. Η κυρία Μορβάη μας είπε ότι δεν λειτουργεί η συνεργασία. Είναι πολύ εύκολο να φέρνει κανείς παραδείγματα. Φυσικά, είναι πολύ δραματικές οι περιπτώσεις που αναφέρατε. Δεν θα διαφωνήσω με το δράμα των παιδιών. Αλλά ε, δεν αρκεί να αναφέρουμε δύο-τρία δραματικά περιστατικά για να πούμε ότι δεν λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αυτός τρόπος να παρουσιάζουμε τα πράγματα. Εγώ μπορώ να φέρω τρία παραδείγματα όπου όλα λειτουργήσαν τέλεια και η συνεργασία υπήρξε τέλεια και ότι όλα ήταν υπέροχα. Επομένως δεν είναι σωστό να προσεγγίζουμε το θέμα με αυτόν τον τρόπο. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Κύριε Μούλντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά μπορούν να υποθούν για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Αλλά καλό είναι να υπάρχει ένας κοινό χώρος όπου να τυχάνουν προστασίας οι πολίτες και να υπάρχει ένας κοινό νόμος και γι' αυτό νομίζω ότι αναπόφευκτα θα έπρεπε να υπάρχει ένας Ευρωπαίος εισαγγελέα. και το περιμένουμε αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιμένουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Δεύτερο ε, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ε, αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορες συζητήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας για, για την προστασία των δεδομένων. Μιλούμε ίσως για κάποιον κανονισμό, για την, τις τεχνικές πρόοδους, τις πρόοδους, τις τεχνολογίες που είναι τόσο γρήγορες, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθούμε. Αλλά πρέπει να το προσπαθήσουμε. Τώρα για την ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Έχουν, έχουν γίνει προσπάθειες στο πλαίσιο του SWIFT και των, του PNR και ξέρω ότι δίνουμε πολλές πληροφορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσαμε τις ίδιες πληροφορίες για Αμερικανούς πολίτες, θα το ενέκρινε αυτό το Κογκρέσο, θα τις έδινε στην Ευρώπη. πούμε ότι είναι πληροφόρηση από τη μία πλευρά και μόνο. Πρέπει να, να δούμε τις πληροφορίες που έχουμε από δικά μας στοιχεία για το SWIFT και το PNR, για τους καταλόγους επιβατών και χρειάζεται να το εξετάσουμε αυτό. Υπάρχουν επίσης προτάσεις για τη μετανάστευση, για το πακέτο Σέγγεν κλπ. Αλλά την ενσωμάτωση και ένταξη δεν έχουμε εξετάσει βάθος και νομίζω ότι είναι όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν ξέρω ε, αν θα μπορούσαμε να έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία, μάλλον δεν μπορούμε, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να διδαχθούμε ημένα από τους δε. Να είναι μια αξιολόγηση ομοτήμων. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Λάμπερτ. Θέλετε να συμβάλλετε στη συζήτηση, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη που έφτασα αργά, απλά συμμετείχα σε μια ψηφοφορία σε άλλη επιτροπή. Ε, να απαντήσω, να σχολιάσω ένα-δυο πράγματα που υπόθηκαν ε, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση ή την έλλειψή της. Το ένα από τα σχόλιά μου έχει να κάνει με το ζήτημα των δεδομένων φυσικά. Τι κάνουμε με τα προγράμματα επίβλεψης και εποπτείας των φορέων που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Έχουμε διάφορους φορείς για αυτά, αλλά ίσως ε, δεν εκμεταλλευόμαστε σωστά τη δουλειά τους ή δεν βλέπουμε πώς εναρμονίζονται σωστά με δουλειά που γίνεται σε άλλους τομείς. Σε σχέση με τη διάσταση της ενοποίησης, της ένταξης, έχουμε το Ταμείο Ένταξης, πρόσφατα είχαμε και μια έκθεση με την Επιτροπή Απασχόλησης ε, για το θέμα της ένταξης στην αγορά εργασίας αλλά νομίζω ότι λείπει ένα άλλο στοιχείο από τη συζήτηση για την μετανάστευση. Είναι η εγκατάσταση και δεν εννοώ η μετεκατάσταση των προσφύγων, γιατί εκεί έχει γίνει κάποια πρόοδος, αλλά εξακολουθούμε πάντοτε να κοιτούμε το ζήτημα της μετανάστευσης σαν να πρόκειται για κάτι βραχυπρόθεσμο. Είναι ένα από τα στοιχεία που λιγότερο έχουμε συζητήσει, γιατί υπάρχουν διάφορα κενά μεταξύ των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας και δεν είναι σαφές πώς διαπλέκεται το ένα με το άλλο και ποια είναι η κατάσταση η οποία τελικά διαμορφώνεται και ισχύει. Ευχαριστώ, κυρία Λάμπερτ. Ε, από ό,τι βλέπω θα ήθελε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετέχει στη συζήτηση. Υπάρχει ένας... η κυρία Σιπάλα ε, θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Αλλά υπάρχει και εκπρόσωπος από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, καταρχήν ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χαιρόμαστε με την απόφαση της Επιτροπής σας να ετοιμάσει μια έκθεση για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και να φέρει και κάποιες ιδέες για το μέλλον θεωρούμε ότι θα είναι πολύ χρήσιμη η έκθεση αυτή για την συζήτηση της μελλοντικής ε, εξέλιξης ε, των εσωτερικών και θα αξιολογηθ... μια προσπάθεια που θα αξιολογήσει τις μέχρι τώρα επιτυχίας και θα διαπιστώσει τι ακόμα λείπει. Ε, με την κυρία Ρέντινγκ και με την κυρία Μάλστρομ έχει γίνει μια συζήτηση που έχει προσφέρει πολλά στοιχεία. Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποια θετικά θέματα. Θέλω να τονίσω ορισμένα. Θα υπάρξει η συγκεκριμενοποίηση και η υλοποίηση ενός στόχου και συγκεκριμένα ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα. Η οδηγία για την ενιαία άδεια οδήγησης που θα απλοποιήσει αρκετά τις διαδικασίες, επίσης στον τομέα της εμπορίας ανθρωπίνων όντων και στην εκμετάλλευση των παιδιών. Θέλω να τονίσω επίσης <clears throat> κάποια θέματα στα οποία αναμένεται πρόοδος. Δύο προτάσεις που παρουσίασε η Επιτροπή ήδη από το 2010 και δεν θέλουμε να γιορτάσουμε και την τρίτη επέτειο των διαπραγματεύσεων. Πρόκειται για τους εποχιακούς εργαζόμενους και για τις ε, ε, τεχνολογίες ε, πληροφορικής και επικοινωνιών. Θα θέλαμε... Το ICT δεν είναι ένα κλασικό εργαλείο. Θέλουμε να οξύνουμε τη λειτουργία θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ανταγωνισμού και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Θέλουμε επίσης να βελτιώσουμε την ικανότητα Ευρώπης να προσελκύει ταλέντα ε, στην Ευρώπη. Θέλω να τονίσω επίσης την επιτακτική ανάγκη να επιτευχθεί πρόοδος στο θέμα της δίμευσης των περιουσιακών στοιχείων, αποτελεσματικό εργαλείο καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Χρειάζονται να γίνουν κι άλλα για τους στόχους του προγράμματος της Στοκχόλμης ε, και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και πρόοδος πάνω στην πρόταση για την Europol, ε, την οποία, για την, οποία όλοι περίμεναν με ανυπομονησία και που θα μπορέσει ίσως να υιοθετηθεί πριν από τις επόμενες εκλογές και θα ολοκληρώσω με κάποια πράγματα για το μέλλον. Από τη μια πλευρά θα έχουμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την άλλη χρειάζεται φυσικά και μια στρατηγική ε, να σκεφτούμε τι θα ακολουθήσει το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Ε, στο νου έρχεται το ζωτικό ζήτημα του νέου πλαισίου της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, που είναι ένα θέμα που όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε Δεύτερον, αν θέλουμε πραγματικά να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την προσέγγιση ενός καταλόγου πρωτοβουλειών ή αν θα έχουμε μία πιο ενοποιημένη στρατηγική, πιο συνολική στρατηγική. Και τρίτον, εάν το καθεστώς μετά τη Στοκχόλμη ε, θα είναι μία προσέγγιση ε, συνεργασίας μεταξύ της Κομισιόν, του Κοινοβουλίου και των οργανώσεων ε, της κοινωνίας και όχι μόνο κάτι μεταξύ όχι ένα διάβημα που περιορίζεται μεταξύ των τριών οργάνων. Και τώρα από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τη δουλειά που κάνει, καθώς και τις άλλες δύο επιτροπές και θέλω να πω ότι συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε η προλαλή σας συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας απασχολεί πάρα πολύ η κατάσταση μετά τη Στοκχόλμη, τι θα ακολουθήσει. Υπάρχουν οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, τον διαφορετικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το γεγονός ότι η πολιτική δικαιοσύνης αποτελεί τώρα κανονικά μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, το, το μόνο ερώτημα που τίθεται είναι τι είδους πρόοδος έχει επιτευχθεί ε, τα πέντε τελευταία χρόνια και τι θα γίνει μετά τη Στοκχόλμη. Πάρα πολλές πρωτοβουλίες ε, που δεν έχουν τύχει κατάλληλης ανταπόκρισης. Αυτό μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες. Πολύ καλή συζήτηση. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Γιατί μετά από αυτή τη συζήτηση θα ληφθούν υπόψη όλες οι προσεγγίσεις, τις έχω σημειώσει, για να καταλήξουμε στο τι θα γίνει το επόμενο στάδιο της συζήτησης. Θα πρέπει μαζί με τους συνεισηγητές από τη Γιούρη και την ΑΦΚΟ να κάνουμε τη σύνταξη του εγγράφου που θα υποβληθεί στις Επιτροπές εν ευθέτω χρόνο. θα κάνουμε μια κοινή συνάντηση με τη Γιούρη και την ΑΦΚΟ γύρω στις 9 με 10 Ιουλίου. Θα εξετάσουμε λοιπόν τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε εκ παραλίλου, εμείς και οι άλλες εμπλεκόμενες επιτροπές, Γιούρι και Ιάφκο. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτή τη συζήτηση. Και τώρα ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για το σημείο αυτό και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο. Μου λέει όμως η γραμματεία ότι ο εισηγητής για το επόμενο σημείο δεν είναι ακόμη στην αίθουσα. διότι εμείς ολοκληρώσαμε τα προηγούμενα σημεία 10 λεπτά νωρίτερα. Ας κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα 10 λεπτών και θα επανέλθουμε για το επόμενο σημείο. Ευχαριστώ. Ε?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 I'm ε, ζητώ συγγνώμη, συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Είμαστε παγιδευμένοι εδώ πέρα. Σε αυτό το χώρο της, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που, είναι, δεν συνδέεται τόσο ικανοποιητικά με όλους τους υπόλοιπους. Ε, ε, και δεν μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε το διάλειμμα, αλλά δεν έχει καταφτάσει ακόμη η συγγήτριά μας για το τελευταίο σημείο της μέρης Είναι καθοδόν, αλλά έχει παγιδευτεί και εκείνη σε κάποια άλλη επιτροπή, τη Γιούρη. Καλό θα ήταν να προχωρήσουμε λοιπόν σημείο 13 για την είσοδο και διαμονή ε, πολιτών ε, τρίτων χωρών ε, ε, για την ανταλλαγή φοιτητών, εθελοντική εργασία, έμισθη, άμισθη, πρακτική άσκηση και το καθεξής. Ε, αυτό είναι το θέμα της κυρίας Βίκστρομ. Μπορώ να δώσω το λόγο στον κύριο Μέλτερ. Πότε κατάλαβα ε, είστε διαθετημένος να παρουσιάσετε το θέμα, να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποια στιγμή θα καταφτάσει και η κυρία Βίξτρομ και φυσικά θα ολοκληρώσει τη διοίκηση που θα έχετε αρχίσει εσείς. Ε, σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Σεσίλια μου έδωσε σημειώσεις ε, και θα σας τις διαβάσω με ιδιαίτερη προσοχή. Όταν λέω είμαι τη άποψη, δεν είναι η δική μου άποψη, είναι τη Εσίλια, έτσι, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Αρχίζω. Ε, χαίρομαι που διορίστηκα εισηγήτρια για αυτό το ζήτημα. Πιστεύω ότι πολλά μπορούν να γίνουν για την ε, μετανάστευση στον τομέα της εργασίας ε, και έχουμε σημαντικά καθήκοντα που μας περιμένουν. Ελπίζω σύντομα να βρούμε συμβαστικές λύσεις για την οδηγία για την επιχειρησιακή μετάθεση και για τους εποχικούς εργαζόμενους. Εγώ πιστεύω και ελπίζω ότι ε, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δεν θα είναι τόσο περίπλοκα όπως στο παρελθόν και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και ενδεχομένω να ολοκληρώσουμε αυτή την εργασία μέχρι το πέρα τη τρέχουσα θητεία. Καλωσορίζω την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από ό,τι κατάλαβα, δεν προβλεπόταν στο αρχικό πρόγραμμα εργασία τη. Ε, και προσετέθη στη συνέχεια. Καλωσορίζουμε την προσθήκη αυτή, κυρίως επειδή αφορά ε, πολλούς νέους ανθρώπους. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους αυτής της οδηγίας, ε, μπορούμε να τον εντοπίσουμε στον, ε, στην ευελτίωση των συνθήκων εισδοχής και διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγνώρισης και άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε και ρήτρες διασφάλειες για την προστασία των όλων όσων έρχονται εδώ για να συμβάλλουν στις κοινωνίες μας. Ε, οι φοιτητές και οι ερευνητές ε, μπορούν πλέον να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 12 ε, μήνες μετά την λήξη της σύμβασής τους ή τη λήξη της φοιτησής σε κάποιο πανεπιστήμιο για να μπορέσουν να βρουν μια θέση απασχόλησης. Πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό να τους δώσουμε τη δυνατότητα να διαμείνουν εδώ και να συμβάλλουν στην κοινωνία μας. Η ελευθερία μετακίνηση πρέπει να εφαρμόζεται και σε όσους έρχονται έξωθεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορέσουμε να τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα να παραμείνουν εφόσον έχουν εισέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλες κατηγορίες όπως η άμυστη και η έμυστη, η πρακτική άσκηση καθώς και η ε, έμυστη εσωτερική ε, βοηθή ε, θα συμπεριληφθούν. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε διαφορετικά δικαιώματα σε όλες τις διαφορετικές κατηγορίες και να ανοίξουμε τα μάτια μας και να συνειδητοποιήσουμε ότι μας λείπουν εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευση ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της γύρανσης του πληθυσμού. Χρειαζόμαστε τέτοιους εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευση ταυτόχρονα έχουμε και πολλούς ανέργους και περιπλέκεται η κατάσταση, περιπλέκεται δε τι περιττέρω διότι αν θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και πολίτε τρίτων χωρών. Κάναμε μια... Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η πρώτη σύσκεψη σκιωδών εισηγητών και προσβλέπω στη συζήτηση για να ακούσω τα σχόλια και τι παρατηρήσει των συναδέλφων. Επίση, περιμένω μια ανυπομονησία τη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή και στη συνεργασία ε, με την Ιρλανδική Προεδρία, καθώ και όλε τι επερχόμενε. Ελπίζω ότι όλα τα θεσμικά όργανα θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια τους ώστε να έχουν μια ομαλή ε, προσέγγιση για αυτό το ζήτημα. Επίσης, να σας πω ότι παρότι θα διοργανωθεί την επόμενη εβδομάδα ακρόαση από την Επιτροπή μας στις 5 Ιουνίου από τις 9 ε, μέχρι τις 12.30 στην αίθουσα 5Β1 για αυτό το ζήτημα και σας καλωσορίζουμε όλους σε αυτή την ακρόαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ωραία, σας ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. κυρία Σμιτ, μπορείτε να μας κάνετε μία αναφορά για την έκθεση αυτή. Ναι, ναι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω την πρότασή μας ε, σήμερα. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για το γυναικότερο πλαίσιο. Υπάρχουν πολλοί νέοι άνθρωποι που ε, εκμεταλλεύονται αυτή την ευκαιρία και προσωρινά μετικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις σπουδές τους, ε, ως, για εθελοντική εργασία, ως εσωτερική άμυστη βοηθή και αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες. Η μετανάστευση από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια πηγή ε, εργατικού προσωπικού υψηλής ε, ειδίκευσης, επίσης φοιτητές και ερευνητές από αυτές τις χώρες ε, είναι κατηγορίες ε, ανθρώπων που ε, χρειαζόμαστε όλο ένα και περισσότερο διότι στην παγκοσμιοποιημένη σημερινή οικονομία δεν είμαστε οι μόνοι που προσπαθούμε να προσελκύσουμε ταλαντούχους και ταλαντούχες και άλλες χώρες τώρα τροποποιούν ή πρόκειται να τροποποιήσουν τους όρους εισδοχής των φοιτητών και των ερευνητών για να προσελκύσουν ακριβώς αυτά τα λαμπρά μυαλά. Δεν προτείνουμε κάτι εντελώς νέο. Έχουμε δύο οδηγίες, μία για τους ερευνητές και μία για τους ε, φοιτητές, μαθητές και εθελοντές και άμυστος ε, ασκούμενους. Ε, τώρα προτείνουμε να συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες και θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξεκινούμε εκ του από το μηδέν γιατί καθυστερήσαμε με αυτή την πρόταση. Ε, στο πρόγραμμα δράσης ε, της νόμης μετανάστευσης αρχικά δεν είχε συμπεριληφθεί αυτή η πρόταση, όμως είχαμε την έκθεση υλοποίηση το 2011, από την οποία προκύπτει ότι ε, ανακύπτουν δυσκολίες για την εισδοχή αυτών των κατηγοριών μεταναστών. Ξέρουμε επίσης ότι έχουν αλλάξει και οι ίδιες οι συνθήκες σε σχέση με το 2013, παραδείγματο χάρη, μετά την Αραβική Άνοιξη, εφάνει ότι η ανταλλαγή ε, νέων ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να, ε, είναι κάτι που πρέπει να συμβαίνει σε σχέση με τις γειτονικέ μας χώρες. Μην ξεχνούμε επίσης ότι η κυκλοφορία εγκεφάλων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να αναβαθμίσει σχέσεις μας με τρίτες χώρες. Εξού και η αναθεώρηση και η κωδικοποίηση ε, ε, και ομαδοποίηση άλλων οδηγιών και κατηγοριών που έχουν παρεμφερεί προβλήματα και ε, άρα είναι παρεμφερείς και εφαρμοστεί οι κανόνες. απλούστευση λοιπόν και ενισχυμένη διαφάνεια. Αυτή είναι η δύο βασικοί στόχοι. Τι θα αλλάξει τώρα με αυτή την πρόταση. Πρώτα απ' όλα υπήκοοι τρίτων χωρών που ε, διαμένουν ε, μέχρι τους τρεις μήνες ή πάνω από τρεις μήνες ε, και είναι εφαρμοστή η διάταξη για τις θεωρήσεις. Οι επιπρόσθετες κατηγορίες, έμισθη και άμισθη εσωτερική βοηθή δεν καλύπτονται αυτές τις δύο κατηγορίες από την κειμένη νομοθεσία, όμως έχουν παρεμφέρει προβλήματα, κυρίως χρειάζονται προστασία διότι βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και ενδέχεται να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης. Η πρόταση για τους εποχιακούς εργαζόμενους δεν είναι μια πρόταση μόνο για την εισδοχή τους, αλλά ένας άλλος στόχος της πρότασης είναι η αποφυγή ακριβώς της εκμετάλλευσης και η παροχή βοήθειας και προστασίας. Αυτό ισχύει και για τους εσωτερικούς άμεστους βοηθούς Το δεύτερο σημείο που θα αλλάξει είναι ότι θα δεσπίσουμε κανόνες για μαθητές, για εθελοντές και για άμυστους ασκούμενους. Θα είναι υποχρεωτικές και όχι πλέον προαιρετικές ε, αυτές οι διατάξεις και οι οργανώσεις που αναλαμβάνουν την ανταλλογή εθελοντών και ε, μάθητων αντιμετωπίζουν προβλήματα ακριβώς λόγω της διαφοράς των εφαρμοστέων διατάξεων κράτος μέλος. Και όπως σας είπα, ε, καλύπτουμε τώρα, ε, πλέον θα καλύπτουμε μάλλον και τους άμυστους ασκούμενους. Τέλος, ε, για όλες αυτές τις κατηγορίες θα έχουμε σαφέστερες διευκρινήσεις ως προς την εισδοχή τους θα είναι διαφανέστερη και απλούστερη η διαδικασία και οι κανόνες που θα εφαρμόζονται για την άδεια διαμονής αλλά και για τη θεώρηση, διότι οι φοιτητές και ερευνητέ ένα βασικό πρόβλημα που έχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι πληρούν όλους τους όρους εισδοχής, έχουν την άδεια αλλά δεν λαμβάνουν τελικά τη θεώρηση και δεν μπορούν να εισέλθουν στη χώρα. Ε, οπότε με την οδηγία αυτή ο στόχος μας είναι να ρυθμίσουμε αυτό το ειδικό πρόβλημα. Ε, από διαδικαστικής πλευράς θα υπάρχουν ε, εχέγγυα και ρήτρες διασφάλισης, ε, χρονικός περιορισμός 60 ημερών για να απαντήσουν οι αρμόδιες αρχές και μπορεί να μειωθεί αυτό και σε 30 ημέρες ε, για όλους όσους έρχονται με το Erasmus Mundus ή με το Marie Curie Fellowship, τέτοια πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να προαγάγουμε επίσης την κινητικότητα στο ιστορικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κινητικότητα των φοιτητών, των ερευνητών, των μελών ε, το, της οικογένειας τους ε, και των έμιστων ε, ασκούμενων με τρόπο ώστε να μετακινούνται ελεύθερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε επίσης σαφέστερους κανόνες, όπως σας είπα για τους ερευνητές Marie Curie και τους φοιτητές του Erasmus Mundus, η θεώρηση που θα εκδίδεται στο πρώτο κράτος μέλος θα ε, ισχύει και σε άλλα ε, κράτη, αν έχει δηλωθεί αυτό εξ αρχής. Τέλος, ε, πρόσβαση στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι φοιτητές μπορούν να εργάζονται για τουλάχιστον 10 ώρες την εβδομάδα. Τώρα θα ανέβει αυτό το όριο στις 20 ώρες εβδομαδιαίως. Έτσι μπορούν ε, να, ε, όχι μόνο να εξασφαλίζουν τα προστοζήρα, αλλά και να συμβάλλουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον προπολογισμό της Ένωσης. Ε, κατόπιν ε, οι φοιτητέ μετά το πέρας ε, των σπουδών τους, οι ερευνητές μετά το πέρας σύμβασής τους θα μπορέσουν να παραμείνουν 12 μήνες για να συνεχίσουν τις σπουδές ή να ιδρύσουν επιχείρηση βάσει πολύ συγκεκριμένων διατάξεων που προσδιορίζονται στην πρόταση. Αυτό δεν σε ισοδυναμεί με αυτόματη πρόσβαση στην αγορά εργασίας γιατί υπάρχει και η εθνική άδεια εργασία που παραμένει η εθνική αρμοδιότητα αλλά τουλάχιστον οι φοιτητέ και οι ερευνητέ θα μπορέσουν να παραμείνουν στην επικράτεια του κράτου για να μην χάσουμε αυτά τα ταλέντα που αποκτήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άνθρωποι που ήδη γνωρίζουν τη γλώσσα και έχουν δεξιότητες που είναι ήδη αναγνωρισμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι απέκτησαν ακριβώς αυτές τις δεξιότητες στην Ένωση. Τέλος, σε πιο προκεγορημένα δικαιώματα για αυτές τις κατηγορίες... Ε, Ε, θέλουμε με αυτή την πρόταση να καλύψουμε τα νομικά κενά, να προσελκύσουμε ταλαντούχου υπηκόου ε, τρίτων χωρών, να τονώσουμε την ανάπτυξη και την ε, καινοτομία, και να έχουμε μια πραγματικά ε, ε αμοιβαίως ε, ε, εποφελή ανταλλαγή ταλέντων και θα συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρος. Εμείς σας ευχαριστούμε. Τώρα θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία και στην Ιρλανδική Προεδρία να μας ε, να εκφράσει την άποψή της. Κύριε Ρότουαρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και τη θέση του Συμβουλίου και να σας δώσουμε μια γενική εικόνα για ε, την θέση που ακολουθεί το Συμβούλιο. η Ιρλανδική Προεδρία προσπαθεί να βρει κάποια συμβιβαστική πορεία και κάποια συμφωνία για τις δύο αυτές οδηγίες και θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για να επιτευχθεί η πρόοδος για τη νέα οδηγία γιατί πολλές διατάξεις ε, μπορούν να επαναληφθούν και στη νέα οδηγία εφόσον έχουμε και τη, τη συμφωνία του Κοινοβουλίου σε ορισμένε διατάξεις. Σε σχέση με τη νέα οδηγία, το Συμβούλιο χαιρετίζει την οδηγία δεδομένης της προστιθέμενης αξίας ε, που θα φέρουν ε, τα πρόσωπα αυτά ε, στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό αυτή τη στιγμή. Η Ιρλανδική Προεδρία θέλει να δείξει τη δέσμευσή της για την επιτυχία προόδου και ήδη μέσα σε τέσσερις εβδομάδες αρχίσαμε την ανάγνωση που ελπίζουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί επί Ιρλανδικής Προεδρίας. Έχουν γίνει ήδη δύο συνεδριάσεις στο Συμβούλιο και ε, θα γίνει και άλλη συνάντηση των εμπειρογνωμόνων πριν το τέλος της ελληνικής προεδρίας. Η συνάδελφος εξ αριστερών εκπροσωπεί την ε, Λιθουανική Προεδρία που ήδη έχει προγραμματίσει πέντε μονοήμερες συναντήσεις για τη συζήτηση αυτού θέματος. Άρα το Συμβούλιο δεν ε, θα κολλησιεργήσει καθόλου, θα συζητηθούν και σε υψηλό επίπεδο στη Σκύφα αρχές Ιουλίου. Βλέπετε λοιπόν ότι το Συμβούλιο σαφώς έχει αναλάβει δέσμευση και η Ιρλανδική Προεδρία και η επόμενη Λιθουανική Προεδρία ε, έχουν δεσμευτεί ότι θα γίνει πρόοδο στο θέμα αυτό. Το Συμβούλιο λοιπόν ε, θα συνεχίσει την ε, πορεία και ελπίζουμε όσο συνεχίζουμε εμείς τη συζήτηση να ληφθούν υπόψη αυτά τα θέματα και σε άλλα επίπεδα. Περιμένουμε και τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου και θα είμαστε πια σε καλή θέση για να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσει, να αρχίσει μάλλον η Λιθουανική Προεδρία διαπραγματεύσεις για πιθανή συμβαστική λύση ώστε να επιτύχουμε συμφωνία για το θέμα αυτό. Από την πλευρά του Συμβουλίου θέλω να πω ότι χαιρετίζουμε την οδηγία και τα ωφέλη από τέτοιες διατάξεις για τα άτομα αυτά που έρχονται να εργαστούν και να ζήσουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά το Συμβούλιο έχει κάποιες ε, ανησυχίες για κάποιες υποχρεωτικές διατάξεις σε ορισμένους τομείς. Για για τους ε, άμυστους βοηθούς ΟΠΕΡ, για τους άμυστους καταρτιζόμενους, ε, μαθητές σε ανταλλαγές κλπ. Ίσως κάποιες από αυτές τις υποχρεωτικές διατάξεις να πρέπει κάπως να αποδυναμωθούν, αλλά θα είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση για τα θέματα αυτά. Όσον αφορά τις υποχρεωτικές διατάξεις είτε για τους ερευνητές, είτε για τους μαθητές, είτε για τους άμυστους, εσωτερικούς άμυστους βοηθούς, θα, θα χρειαστούν και κάποιες ε, ρήτρες διασφάλισης για το Συμβούλιο για να μην υπάρξει κατάχρηση αυτών των διατάξεων. Ε, πιστεύουμε ότι καμία από τις οδηγίες αυτές, ε, ούτε αυτή ούτε για τους ICT, θα πρέπει να αφήσει ε, το ενδεχόμενο κατάχρησης αυτών των διατάξεων, ε, ώστε να έχουμε παράνομη μετανάστευση. Κλείνοντας λοιπόν, εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με τους συνομοθέτες μας για να επιτύχουμε κοινή πρόοδο για το θέμα αυτό. Ήδη έχουμε κάνει δύο συνεδριάσεις με την εισηγήτρια, την κυρία Βίξτρομ, η οποία δείχνει ιδιαίτερα θετικό πνεύμα για να επιτύχουμε πρόοδο και συνεργαζόμαστε και μαζί της και οι συνάδελφοι από τη Λιθουανική Προεδρία θα συνεχίσουν να συνεργάζονται μαζί της για να επιτύχουμε το συντομότερο δυνατό κάποια πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την Επιτροπή, ακούσαμε το Συμβούλιο. Και μια και η κυρία Βίξτρομ δεν είναι παρούσα, ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Κοέλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και ο κύριος Μόλτερ, έτσι και εγώ Έχω τις σημειώσεις της κυρίας Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλτ που θα είναι σκιώδη συγγήτρια από το ΕΛΚ. Μου ζήτησε να σας μεταφέρω τα έξη. Ως σκιώδη συγγήτρια από το ΕΛΚ, εγώ, εγώ ως Άννα Μαρία Κορέτσα Μπίλτ δηλαδή, χαιρετίζω την πρόταση της Επιτροπής για την ε, αποδοχή υπηκών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκοπό των σπουδών, ανταλλαγών ε, κλπ. Για τον, να επιτρέψουμε σε ερευνητές και μαθητές να φέρουν τις δεξιότητες και ικανότητές τους στην Ευρώπη ε, θα δώσουμε τη δυνατότητα σε ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καινοτομία στην έρευνα στην Ευρώπη. Κάτι το οποίο είναι απολύτω απαραίτητο για να γίνει πιο ανταγωνιστική η Ευρώπη. Το να θέσουμε κοινού κανόνε σε αυτό το τομέα είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να επωφεληθούμε από τέτοιου είδου μετανάστευση και ταυτόχρονα να δώσουμε δίκαιη μεταχείριση και ρήτρε διασφάλιση για αυτέ τι ομάδε υπηκών τρίτων χωρών που έρχονται να ζήσουν και να εργαστούν στην Ευρώπη για κάποιο χρονικό διάστημα. Η κυρία Κοράζα Μπίλκ λοιπόν προσβλέπει στην συζήτηση των θεμάτων αυτών με την εισηγήτρια και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτό το μέτρο θα εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για αυτούς που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για σπουδές και έρευνα, κατά τρόπον ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και συμβατότητα με τις εθνικές νομοθεσίες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, κυρία Φλότχ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα συμφωνήσω με αυτά τα οποία μέχρι τώρα ελέγχθησαν. Να χαιρετίζω την πρόταση αυτή. Θεωρώ και εγώ ότι είναι πολύ θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει αυτό το κείμενο. Είναι ένα θετικό μήνυμα για την κινητικότητα των νέων και των όχι και τόσο νέων. Υπάρχει ένα συμφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διακίνηση αυτών των ατόμων, ιδεών, γνώσεων, με προοπτικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Πολύ θετικά όλα αυτά. Τα άτομα αυτά και με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής Μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν πολλά εμπόδια. Υπήρχε περιοριστική πολιτική για τις θεωρήσεις διαβατηρίου, οικονομικές δυσκολίες, δυσκολίες στέγασης κλπ. κλπ. Όλες αυτές οι δυσκολίες πρόσβαση στην αγορά εργασίας και για το θέμα αυτό το ερώτημα που τίθεται είναι το αν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα τελικά αρκετά ελκυστικό για τους ερευνητές, για τους φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευόμενους και άμυστους εσωτερικούς βοηθούς, ούτως ώστε να συνεχίσουν να κυκλοφορούν οι ιδέες και οι γνώσεις και να εμπλουτίζουν την ευρωπαϊκή κοινωνία και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι η πρόταση αυτή ανταποκρίνεται σε πολλά σημαντικά ερωτήματα. Μπορούμε να βελτιώσουμε το θέμα των θεωρήσεων διαβατηρίου, παραδείγματο χάρη. Ένα άτομο που είναι γεγραμμένος σε έναν οργανισμό ή ένας ερευνητής που έχει μια σύμβαση με ένα ερευνητικό φορέα, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να παρεμποδιστεί στο να έχει πρόσβαση με περιορισμούς θεώρησης διαβατηρίου κατά κανένα τρόπο δεν πρέπει η θεώρηση διαβατηρίου να αποτελέσει εμπόδιο για τέτοιου είδου ερευνητέ. σω να πρέπει εδώ να γίνουμε πιο ξεκάθαροι και πιο συγκεκριμένοι. Ε, πρέπει να αφήσουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα του να μειώσουν την πρόσβαση των φοιτητών σε κάποιε μορφέ απασχόληση ανάλογα με την ε, αγορά και τον κλάδο εργασία. Α το σκεφτούν αυτό οι εισηγητέ. για τους φοιτητές η εργασία θα είναι το βασικό μέσο χρηματοδότησης των σπουδών τους και αυτό μπορεί να κάνει ελκυστική την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως πρέπει και να διευκρινίσουμε για τις θεωρήσεις διαβατηρίου ότι εξ αρχής θα πρέπει να υπάρξει κάποια εγγύηση πολλαπλών εισόδων για τις θεωρήσεις διαβατηρίου, επαναλαμβάνω, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα κάποια στιγμή. Και όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, 12 μήνες ε, με κάποια ε, αυτή απόδειξη ότι αναζητούν εργασία και μετά από 6 μήνες να έχουν κάποια δυνατότητα πρόσληψης αναλόγως των περιστάσεων. Ίσως αυτές οι προθεσμίες είναι λίγο σφιχτές. Ε, δεν ξέρω πώς έπρεπε να λέμε 6 και 9 μήνες αντί 3 και 6 μήνες. Άλλο ένα θέμα προς εξέταση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας και την ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά το κόστος, ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ίση μεταχείριση και να φροντίσουμε τα κράτη-μέλη, αφού περάσει σε εθνικό δίκτυο να, να φροντίσουν τα κράτη-μέλη να δίδουν σαφή ενημέρωση επί της διαδικασίας, διαδικασία που είπαμε θα έχει γίνει ελκυστική, ούτω ώστε αυτή η πρόταση να αλλάζει την κατάσταση. Φέτος η Γαλλία είναι πέμπτη στη σειρά μεταξύ ελκυστικών χωρών. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πλέον ελκυστική χώρα με 400.000 φοιτητέ. Ε, η Αυστραλία όμως έχασε τη ε, πήρε τη θέση της Γαλλίας και έτσι έχει χάσει η Γαλλία μια θέση. Άρα χάνουμε ανταγωνιστικότητα διεθνώς. Και άρα είναι πολύ σημαντικό με μια τέτοια πρόταση να μπορέσουμε να είμαστε πιστικοί και ελκυστικοί για τους μαθητές, φοιτητές, ερευνητές και νέες κατηγορίες που καλύπτονται από την πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν, ευχαριστώ την εισηγήτρια μέσω αυτών που μας μετέφερε ο κ. Μούλντερ. Η συνάδελφος Jean Lambert που ασχολείται με το θέμα αυτό στην Επιτροπή Απασχόλησης μου έδωσε να καταλάβω ότι για τα θέματα των κοινωνικών δικαιωμάτων υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και κάποιες διευκρινήσεις που πρέπει να γίνουν και θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην Επιτροπή Απασχόλησης που θα εξετάσει αυτά τα θέματα εμπεριστατωμένα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία Ματιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ θετικά αντιμετωπίζουμε και εμείς την πρόταση αυτή δεν είναι καινούργια, αλλά είναι πολύ επίκαιρη. Είναι ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να είναι χώρος υποδοχής νέων και νέων ταλέντων. Με την ελπίδα θα τους κρατήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι μεσοπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πρόβλημα όσον αφορά την ε, απασχόληση, αλλά εδώ έχουμε μια πολύ καλή πρόταση με νέα δικαιώματα για τους ερευνητές, για τους φοιτητές, το δικαίωμα παραδείγματο χάρη να μπορούν να εργάζονται σε μερική απασχόληση για να χρηματοδοτήσουν τι σπουδέ του ή να έχουν κάποια κινητικότητα μέσα σε 12 μήνε μετά τι σπουδέ του, ώστε να μπορέσουν ε, να ε, αναζητήσουν εργασία. Κάποιες διατάξεις για την ε, υποδοχή και μελών της οικογένειας, για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τη δυνατότητα για του φοιτητέ να μπορούν για μέγιστο διάστημα έξι μηνών να πάνε και στην άλλο κράτο μέλο. Αυτά είναι πολύ θετικέ προτάσει τη Επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Τριανταφυλλίδη. <coughs> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω και ο εκ μέρου τη ΓΚΟΕ χαίρομαι ιδιαίτερω που έχουμε αυτή την αναδιατύπωση ενώπιών μας και ελπίζω ότι εδώ θα έχουμε σαφή προστιθέμενη αξία για τους ε, μετακινούμενους εργαζομένους και τονίζω ότι οι εταίροι μας και οι γείτονές μας ε, περίμεναν ε, εδώ και καιρό για τέτοιου είδους πρόταση για να διευκολυνθούν οι επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υπάρχουν βέβαια κάποιες αντιφάσεις, γιατί από τη μια πλευρά λέμε ότι θέλουμε στενότερες σχέσεις και καλύτερη συνεννόηση, από την άλλη πλευρά απαιτούμε από αυτούς να διαχειρίζονται τα εξωτερικά μας σύνορα και να σταματούν τις ροέ μετανάστευση ε, χωρίς να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποσπασματική και πολύπλοκη η πολιτική μας για την μετανάστευση. Αντί να έχουμε ένα σαφές πλαίσιο για υπηκόους τρίτων χωρών που θέλουν να έρθουν για σπουδές και εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπίσουμε ένα πολύπλοκο καθεστώς νόμων με πολύπλοκες διαδικασίες και δικαιώματα ανάλογα με τις διάφορες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών. Πιστεύουμε ότι η συνένωση αυτών των κατηγοριών μπορεί να είναι θετικό βήμα εφόσον είναι απλουστευμένες οι διαδικασίες και εφόσον τους χορηγούνται τα απαραίτητα δικαιώματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να αναλύσουμε τις αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή, να διασφαλίσουμε ότι όντως διευκολύνουν και δεν περιορίζουν ε, την ε, κυκλοφορία αυτών των εργαζομένων και αυτών των προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να κάνω και μια προκαταρκτική παρατήρηση για την επιλογή τη διατύπωση που έχουμε σε αυτό το κείμενο, ώστε να δίνουμε το σωστό μήνυμα προ του φίλου και εταίρου. Και ξέρω ότι πολλέ φορέ έχουμε κάνει την ίδια συζήτηση. Πιστεύω όμω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επιμείνουμε ε, να μιλάμε για ε, κανονική regular μετανάστευση και όχι νόμιμη και παράνομη μετανάστευση γιατί η σημασιολογία είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τα δικαιώματα ε, των μεταναστών όπως πολύ συχνά επαναλαμβάνουμε. Η μετανάστευση είναι κάτι το θετικό και όχι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει ποινικό αδίκημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπρόνς. Μιλούσαμε για την εμπορία ανθρώπων προηγουμένως και μιλούσαμε κυρίως για την μεταφορά προσώπων διεθνώς με σκοπό την εκμετάλλευσή τους συνήθως αυτός ο οποίος θίγεται είναι ο μεταφερόμενος, ο διακινούμενος, αλλά θα μπορούσε και η χώρα να πλήττεται, η χώρα από την οποία μεταφέρεται ε, αυτό το άτομο. Βέβαια αυτός που κερδίζει πάντοτε είναι ο διακινητής ανθρώπων. Στην τέταρτη παράγραφο του επεξηγηματικού σημειώματος της Επιτροπής υπάρχει εξή διατύπωση, παραθέτω. Μετανάστευση ε, από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια πηγή ε, ατόμων με υψηλές δεξιότητες. Δεν λέει από ποιες χώρες θα έρθουν, αλλά τέτοιου είδους πρόσωπα έρχονται συνήθως από τις πιο φτωχές χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Ίσως το 2010 να θυμάστε πολλοί από εσά ότι ο πρόεδρος του Μάλι τότε είχε έρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε λάβει το λόγο και ε, είπε ότι η χώρα του που πλήττεται από τη φτώχεια κάνει θυσίες για να εκπαιδεύσει και να καταρτήσει ε, τα ικανά άτομα που υπάρχουν στη χώρα. Όμως αυτοί που, έχουν, που αποκτούν ε, δεξιότητες στον τομέα της ιατρικής ε, ή στον τομέα των επιχειρήσεων πολύ συχνά στρατολογούνται και προσλαμβάνονται για να δουλέψουν στην Ευρώπη ή στη Βόρεια Αμερική αντί να μείνουν στη χώρα. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρώπη έχει μια φτηνή παροχή εργατικών χεριών χωρίς να πληρώσει για την εκπαίδευσή τους. Φέροντα εκπαιδευμένα άτομα από τον τρίτο κόσμο στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν είναι εμπόριο ανθρώπων. Αν δεν είναι εμπόριο ανθρώπων, τι είναι. Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζονται επαγγελματίες ε, υγείας ή ε, ασθενείς ε, και φτωχοί στις τρίτες χώρες. Θεωρούμε ότι μπορούμε εμείς να αλληλετούμε ε, ε, τους εκπαιδευμένους ε, στις χώρες του τρίτου κόσμου για να τους φέρουμε στην Ευρώπη τα νοσοκομεία στην Ευρώπη θα μπορούσαν να προσφέρουν πακέτα εξαποστάσεως εκπαίδευσης και να προσπαθούν με τρόπο οικονομικά αποδεκτό ε, να εκπαιδεύσει και να προσθέσει ε, θετικά στοιχεία σε αυτά τα οποία χρειάζονται οι χώρες του τρίτου κόσμου. Ευχαριστώ πολύ και δίνουμε το λόγο και πάλι στην Επιτροπή για να κλείσει το θέμα, γιατί σήμερα συζητάμε την πρόταση της Επιτροπής. Άρα θα δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή για να κλείσει αυτό το σημείο με την τελική της παρέμβαση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ θετική ανταπόκριση στην αρχική μας παρουσίαση. Ε, προσμένω στη συνεργασία μου με την εισηγήτρια, την κυρία Βίλκστρομ, με την Επιτροπή Γιούρι, που και εκείνη είναι πολύ θετική. Δεν βλέπω να, ανάγκη να απαντηθεί κάτι συγκεκριμένο εδώ. Αναφέρθηκε ο κίνδυνος της κατάχρησης. Έχουμε συμπεριλάβει άρθρα τα οποία προσεγγίζουν το θέμα της κατάχρησης, ε, των καταχρήσεων. Θα το εξηγήσουμε και σε μελλοντικέ μας συναντήσεις. Θα θέλαμε να σας ευχαριστούμε για αυτή τη θετική ανταπόκριση και προσμένουμε με χαρά ε, την ευκαιρία να σας δώσουμε και άλλες εξηγήσει για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αναφέρθηκε η οδηγία για τους εποχιακούς εργαζόμενους και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό μετά από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά με το ε, Κοινοβούλιο και ελπίζουμε και με το Συμβούλιο και ελπίζουμε στις προσεχείς εβδομάδες να καταλήξουμε σε συμφωνία πάνω σε αυτές τις δύο σημαντικές προτάσεις και να βρούμε λίγο περισσότερο χώρο για να, να εμβαθύνουμε περισσότερο, περισσότερο πόσο κάναμε σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες η συζήτηση συνεχίζεται και θα σας κρατήσουμε ενήμερους. Ε, υπάρχει η συνεδρίαση των συντονιστών, η οποία θα είναι και κλεισμένων των θυρών. Ωστόσο, οι περισσότεροι συντονιστές δεν θα τα καταφέρουν να έρθουν εδώ. Ας προχωρήσουμε λοιπόν άμεσα, δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις, μόνο ενημέρωση. Οι συντονιστές να παραμείνουν στην αίθουσα, όλοι οι άλλοι να φύγουν και συνεχίζουμε τις εργασίες της Επιτροπής στις 9 αύριο το πρωί. Please, all of the members who are not allowed to be part of the coordinators meeting, leave the room in silence so that we can proceed the sooner the better. Thank you.